morning, dear colleagues. Let's resume our work. Yesterday we had a... Ας επαναλάβουμε και συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Χθες είχαμε μια, ένα σεμινάριο για την Συμφωνία Ενωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κεφάλαια που αφορούν τις εργασίες της ΛΥΜΠΕ. Αλλά έχουμε και σήμερα το πρωί μια ε, ημερήσια διαταξή, έχοντας υπόψη ότι έχουμε ψηφοφορίες στις 12 παρα 10, 11 και 50. Οπότε πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί με το χρόνο. Θα πρέπει να έρθουν ε, όλοι με τις ηλεκτρονικές τους κάρτες. Και μέχρι τις 12 παρα 10 Ελπίζω ότι θα έχουν έρθει και περισσότεροι βουλευτές στη συνεδρίαση. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να τελειώσουμε στις 12 παρα 10. Να περάσουμε στο σημείο 7, κατάσταση των διαπραγματεύσεων των συμφωνιών επανεισδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ακούσουμε μια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα ακούσουμε και τους συντονιστές και τον εισηγητή και τους σκιώδους εισηγητές για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει γραπτές πληροφορίες για τις ενεξελίξεις διπλωματεύσεις, για τις μελλοντικέ συμφωνίες και για τις υπάρχουσες συμφωνίες επανεισδοχής. Θέλουμε να δούμε τι ε, δηλώσεις και ε, συμφωνίες υπάρχουν με τρίτες χώρες, ακόμα και άτυπες, για τα θέματα αυτά. Θα ακούσουμε λοιπόν την κυρία Παριάτ. Τη συγχαίρουμε παρεμπιπτόντως για τον διορισμό της στην Γενική Διεύθυνση Home, όλα τα μέλη της Επιτροπής μας και σας ευχόμαστε επί τη ευκαιρία καλή τύχη στις νέες σας αρμοδιότητες για τα επόμενα χρόνια. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά για να έχουμε αμέσως μετά χρόνο για συζήτηση. Έχετε το λόγο. Και πάλι συγχαρητήρια. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με καλωσορίζετε σήμερα εδώ. Και ευχαριστώ για τις ευχές σας. Όλοι χρειαζόμαστε σε αυτή τη δουλειά υποστήριξη. Ελπίζω λοιπόν να μας βοηθήσετε να προχωρήσουμε με τα δύσκολα αυτά θέματα. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Κάποια πρόσωπα μου είναι οικεία. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Και επειδή είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι θέλω να έχουμε στενή συνεργασία. Και θα έρχομαι όσο πιο συχνά γίνεται και όποτε χρειάζεται για να συνομιλούμε. Διότι ο στόχος είναι να είμαστε όσο διαφανέστεροι γίνεται στη δουλειά μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας τηρεί ενημερούς. Σήμερα λοιπόν χαίρομαι που μπορούμε να ξεκινήσουμε το διάλογο αυτό με ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα. Ε, επιστροφές Επιστροφέ όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υποχρέωση των χωρών προέλευση να του δεχτούν ξανά. Η εμπειρία μα έχει δείξει ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σφαιρική, μια συνολική αντιμετώπιση των προκλήσεων του φαινομένου της μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μια προσέγγιση η οποία βασίζεται σε κοινέ αξίες και ευθύνες που Πρέπει να αντιμετωπίσουν τα γενεσιουργά αίτια τη παράτυπη μετανάστευση, τη λαθρέα μετανάστευση. Σήμερα 220 κάτι προγράμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προ το καταπίστευμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεπεράσει στο συνολικό ποσό πρικοδότηση στα 4,4 δι ευρώ. Επίση, έχουμε βελτιώσει την διαχείριση της μετανάστευσης, καταπολεμώντας το λαθρεμπόριο και την εμπορία ανθρώπων. Έχουμε σώσει ζωές με 760.000 ανθρώπους να έχουν διασωθεί στη θάλασσα και πάνω από 23.000 μετανάστες στην έρημο, ε, στον Νίγηρα από το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει και εναλλακτικέ λύσει για την λαθρέα μετανάστευση με νόμιμε οδού για μια σειρά από μεταναστευτικού σκοπού, όπω και για την επαναγκατάσταση. Και πάνω από 67.000 ανθρώπου έχουν επαναγκατασταθεί σε κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015. Τέλο, θέλουμε να ασχοληθούμε και με τις ειδικέ ανάγκες όσων έχουν εκτοπιστεί λόγω ένοπλων συγκρούσεων ή διώξεων. Όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει κανένα δικαίωμα για να προστατευτεί διεθνώς ή δεν μπορεί να παραμείνει, πρέπει να επιστρέψει με τρόπο αξιοπρεπή. Για να επιστρέψουν οι παρατύπους διαμένοντες μετανάστευσης πρέπει να έχουμε μια τακτική διαδικασία ασύλου και μετανάστευσης και να είμαστε βέβαιοι ότι τρίτες χώρες συνεργάζονται στις διαδικασίες επανεισδοχής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνεργασία με του ε, παράνομου μετανάστε ή καταστρέφουν τα διαβατήριά του ή τα εγγραφέα του, θα πρέπει οι τρίτε χώρε να ε, μπορούν να εντοπίσουν του προ επιστροφή υπηκόου του και σε αυτό που πρέπει να μπορούμε να υπολογίζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υποχρέωση ε, βάσει του διεθνού δικαίου. Και έτσι δεν υπάρχει πάντοτε ειδική, ανάγκη για ειδική συμφωνία διαθέτηση. Όταν όμω η συνεργασία δεν είναι αρμονική, πρέπει να μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η τρίτη χώρα επιβεβαιώνει την πολιτική της δέσμευση να συνεργαστεί και να συμφωνήσει ε, για κάποια σαφή και ξεκάθαρη διαδικασία. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εγγυάται ότι οι επιστροφές έχουμε μόνο μετά από την προσεκτική εξέταση, την διεξοδική εξέταση κάθε περίπτωσης. Έχουμε μια ξεκάθαρη νομοθεσία και ενωσιακή και εθνική που προβλέπει ε, νομικά εχέγγυα για όλους τους προς επιστροφή ε, ξένους επικόους και σε περίπτωση της μη ε, απομάκρυνσης. Το 2015 είχαμε προτείνει αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για να γίνει αποτελεσματικότερο, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να γίνονται πάντοτε σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε 23 ε, νομικά μέσα επανεισδοχή που ισχύουν και τα οποία διαχειριζόμαστε σε στενή συνεργασία με τρίτε χώρε και κράτη-μέλη. 17 συμφωνίε και 6 ε, διευθετήσει. Όπω ε, θα το πούμε μετά, το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για την επιπλέον συμφωνία με τη Λευκορωσία. Κυρίε και κύριοι, θα είχατε τη δυνατότητα να δείτε τις λεπτομέρειες ε, της επιστολής που σας ε, απέστειλα πρόσφατα για το θέμα αυτό. Και από την τελευταία φορά που συζητήσατε τα θέματα αυτά τον Ιούνιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά κάθε δυνατή ευκαιρία για να ξεκινήσει διάλογο με τις εν λόγω χώρες για τα θέματα της επανεισδοχής. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία νέα συμφωνία, κάποιο νέο μέσο. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε επί τη εφαρμογή των υπαρξών συμφωνιών και διευθετήσεων και έχουμε οργανώσει 22 επιτροπέ ε, για τα θέματα επανεισδοχή και 10 ομάδε εργασία, συνεδριάσει ομάδων εργασία Εν τω σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή των υπαρξών ε, συμφωνιών επανεισδοχή και των ε, σχετικών διευθετήσεων, η συνεργασία με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και δικαιούχους του καθεστώτος απελευθέρωσης θεωρήσεων ή του προενταξιακού συστήματος έχει δώσει καλά αποτελέσματα και έχει τύχει θετική αξιολόγηση από τα μελη Οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, Γεωργία, Αρμενία και Αζερβαϊτζάν, Μολδαβία και Ουκρανία έχουν επίσης σωστά καλά αποτελέσματα επιστροφών τα τελευταία χρόνια. Ενώ τα κράτη-μέλη επιχειρησιακά στα προγράμματά τους δείχνουν ότι υπάρχουν προβλήματα, ε, έχουν βελτιωθεί τα αποτελέσματα. Οι αρχές στη Σρι και στο Κολόμπο έχουν πει ότι έχουν επίσης ε, βελτιωθεί τα ποσοστά επιστροφής και ελπίζουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αρχίσει να λειτουργεί τον Φεβρουάριο θα διευκολύνει την διαχείριση των σχετικών περιπτώσεων Το Πακιστάν επίσης κάποιες φορές ε, αρνείται κάποιες επιστροφές γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκή τεκμηρίωση. Το σύστημα διαχείρισης των επιστροφών όπου έχουν πρόσβαση μόνο τέσσερα με κρατημέλη στην πιλωτική του φάση έχει επιφέρει κάποιες βελτιώσεις. Σήμερα οι ε, συνάδελφοί μου συζητούν με το Πακιστάν μια επέκταση του συστήματος όπου θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλα τα κρατημέλη. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία με την Τουρκία και τη συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία μεταξύ Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ξέρετε, οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι δεν θέλουν να εφαρμόσουν τι διευθετήσει για του επικού τρίτε χώρε και με το καθεστώ απελευθέρωση θεωρήσεων σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή η συνεργασία δεν είναι η ίδια μεταξύ όλων των κρατών μελών και, το, και της Τουρκίας. Επίσης, από το 2016 δεν θέλουν να υπάρξει συνεδρίαση της κοινή Επιτροπής για την Επανεισδοχή, οπότε είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια πολύ τεκμηριωμένη και σαφής αξιολόγηση της συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να επισημαίνει την ανάγκη να εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία σε όλες τις, τις πτυχές και για όλα τα κράτη-μέλη. επειδή αυξάνονται διαρκώς οι αφήξεις μέσω των ε, ελληνικών συνόρων και των ελληνικών νησιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Τουρκία να βελτιώσει τη συνεργασία και να εφαρμόσει το διμερές πρωτόκολλο. Για το πράσινο κροτήρι. Ε, το ποσοστό επιστροφών δείχνει ότι έχει βελτιωθεί η συνεργασία καθώς είναι η μόνη αφρικανική χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνία επανεισδοχής. Η συνεργασία με την Αιθιοπία μετά τι διαδικασίε επανεισδοχή έχει αποδειχθεί δυσχερή στην πρώτη χρονιά εφαρμογή. Όμω οι πολιτικέ δεσμεύσει των αιθιοπικών αρχών για να εφαρμοστούν σωστά οι διαδικασίε ελπίζουμε ότι θα δώσουν σύντομα θετικά αποτελέσματα. Με την ακτή του ελεφαντοστού έχουμε περιορισμένο αριθμό υποθέσεων και τα κράτη-μέλη δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα να βρούμε μια μορφή συνεργασίας. Οι καλές πρακτικές με τη έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα στις συνολικές ε, ε, περιπτώσεις και τα κράτη-μέλη που στο πλαίσιο της συνεργασίας έχουν αποφασίσει να ε, συνεργαστούν, παρόλο που δεν έχουμε πολλές επιστροφές προς τα εκεί. Η Γκάμπια είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Οι καλές πρακτικές για τον εντοπισμό και τις επιστροφέ, ισχύουν από τον Νοέμβριο του 2018. όμω οι αρχές της Γκάμπια αποφάσισαν το Μάρτιο του 2019 να προβλέψουν ένα μορατόριο για όλε τι επιστροφέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω περιορισμού δυνατοτήτων. Η ε, Επιτροπή, η ΕΕ και οι Ευρωπαϊκές Αρχές συνεχίσουν να συνομιλούν με την Κάμπια για να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους. Σε ό,τι αφορά άλλες διευθυντήσεις, για την συνεργασία με το Αφγανιστάν, ο κοινός, ε, η κοινή οδός πρόοδου έχει βελτιώσει τα αποτελέσματα για τις επιστροφές και τις διαδικασίες επανένταξης. Τα κράτη-μέλη συνολικά είναι ικανοποιημένα με την υλοποίηση αυτού της μορφής συνεργασίας. Τέλος, το ποσοστό ε, είναι χαμηλό και αργή, είναι ε, αργή η επεξεργασία και εξέταση των φακελών, όμως τα κράτη-μέλη συνεχίζουν τις προσπάθειές τους και ε, θέλουν να ε, εντείνουν και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα. Τώρα για τις ανεξελίξεις διπλωματεύσεις. Συμφωνίες επανεισδοχής με την Κίνα και ταυτόχρονα συμφωνία διευκόλυνσης θεωρήσεων. Πολύ βραδίως. με την Τινησία και την Νιγηρία. Έχει γίνει πρόοδος το 2018 σε τεχνικό επίπεδο, όμως οι συζητήσεις έχουν σταματήσει για το μεγαλύτερο διάστημα το 2019, γιατί στις χώρες αυτές είχαν εκλογές. Δεν έχουν προγραμματιστεί νέοι γύροι διαπραγματεύσεων από τότε. Οι διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο μπορεί να ξεκινήσουν ξανά στο μέλλον, ως μέλος, μέρος της πολύ στενής συνεργασίας και της στατικικής εταιρικής σχέσης που έχουμε με το Μαρόκο. Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, θα πρέπει οι τρίτες χώρες να συνεχίσουν να συμμετέχουν συστηματικά στις διαπραγματεύσεις και να προσπαθούν να εφαρμόσουν σωστά όλες τους τις πτυχές στη συνέχεια. Αυτό είναι το καθοριστικό μια ε, σωστά εξισορροπημένη εταιρική σχέση είναι η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε τι δυσκολίε διαχείριση τη μετανάστευση και να βελτιωθούν οι συνθήκε και στι χώρε προέλευση. Για να ε, είμαστε βέβαιοι όμω ότι υπάρχει πλήρη συνεργασία από την πλευρά των τρίτων χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει Όπω επανειλημμένως έχει πει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα περασμένα χρόνια, επισημένοντα κυρίως ότι το εμπόριο, η ανάπτυξη και οι συνεργασίες της θεωρήσεις είναι εργαλεία. Ο πρόσφατα αναθεωρημένος κώδικας για τις θεωρήσεις που θα αρχίσει να ισχύει σε λίγες μέρες συνδέει το επίπεδο συνεργασία για τι επανειστοχέ με τρίτε χώρε με την ε, πολιτική έκδοση θεωρήσεων. Αυτό μπορεί να επιτρέψει να υπάρξουν θετικότερα ε, αποτελέσματα και αυστηρότερη εφαρμογή του κώδικα θεωρήσεων ανάλογα με το επίπεδο συνεργασία των άλλων χωρών. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα που ε, είναι ένα ακόμα εργαλείο σε αυτά που ήδη έχουμε ε, και στο φάσμα δικτύων που υπάρχουν για να ενισχυθεί η επανεισδοχή με τις πλατφόρμες για την ηλεκτρονική διαχείριση υποθέσεων, με τους αξιωματικούς συνδέσμους, με τα τεχνικά εργαστήρια για την εκπαίδευση και την κατάρτιση προσωπικού, με την επιχειρησιακή ε, συνεργασία και συμμετοχή σε διαδικασίες επανεισδοχής. Η εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι η διαρκή παρακολούθηση, ο έλεγχο, η επικοινωνία και η στοχευμένη υποστήριξη είναι απαραίτητε για τα εργαλεία επανεισδοχή και προκειμένου να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Όμω πρέπει να δώσουμε και τα σωστά κίνητρα. Η υποστήριξή μα στου επόμενου μήνε, στα πλαίσια τη φερική προσέγγιση για τη διαχείριση τη μετανάστευση, είναι κάτι από αυτά που πρέπει να κάνουμε για να υπάρξει στενή συνεργασία με τι τρίτε χώρε και τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν σωστά τι ισχύουσε συμφωνίε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω ξέρετε, σύντομα θα υποβάλει μια νέα πρόταση για σύμφωνο ε, μετανάστευση και ασύλου και η επανειστοχή θα αποτελεί μέρο του. Ε, θα, πάψω, θα πάψω εδώ και θα είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε ερωτήσει εφόσον έχετε. Το ίδιο και οι συνάδελφοί μου, αν θέλετε περισσότερε λεπτομέρειε γιατί είμαι λίγο καινούρια και προσπάθησα να τα πω όλα, αλλά θα χρειαστώ και τεχνική υποστήριξη. Thank you, We wish you well, but... Uh, Σας ευχαριστούμε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα μέλη που επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστές και μετά από τα υπόλοιπα, με τις παρεμβάσεις των υπολείπων μελών. Να κάνω κι εγώ μια παρατήρηση. Νομίζω κάτι πολύ σημαντικό όταν μιλούμε για επιστροφές και επανεισδοχές. Είναι να μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να αγωνίζεται κανείς για την αλήθεια εναντίον ξεκάθαρα, ξεκάθαρων ψευδών ειδήσεων, ψεμάτων, παραπληροφόρησης, που δεν δημιουργούν μόνο δυσκολίες στην κατανόηση του προβλήματος, αλλά και στη διαχείρισή του. Του ζητήματος μάλλον. Γιατί δεν ισχύει ότι έχει ξεφύγει από τον έλεγχο η μετανάστευση και ότι εισβάλλουν μετανάστες στην Ευρώπη. Έχουν, έχει μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών προς την Ευρώπη. Αυτό που μας λείπει είναι να έχουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα της μετανάστευσης που να είναι ανταξία του ονόματος της. Κάτι που δεν συνέβη ποτέ γιατί μπορεί να έχουμε νομοθεσία και μπορεί να έχουμε ε, νομικά δεσμευτική νομοθεσία όπως για παράδειγμα οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη συνθήκη της Λεσαβόνας για τη δημιουργία του κοινού συστήματος ασύλου, όλα αυτά δεν εφαρμόστηκαν ουσιαστικά στην πράξη ποτέ παρόλα αυτά, ο αριθμός των εισερχομένων μειώνεται και οι επιστροφές είναι περισσότερες από τις παρατυπές εισόδους. Το οποίο στην πράξη σημαίνει ότι κατά τη τιμή και σε ε, σχετικές τιμές ε, η δημογραφική σύσταση της Ευρώπης φθήνει. Και αυτά είναι απλώς στατιστικά στοιχεία απλάς μια πραγματικότητα που θα έπρεπε να μας καθοδηγεί στη συζήτηση για να αποφεύγουμε τη δημαγωγία, το λαϊκισμό και όλα αυτά τα ψέματα που ακούμε για το θέμα. Ας δώσω τώρα το λόγο στους συντονιστές, ξεκινώντας από τον κύριο Λένας που θα εκπροσωπήσει το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε επίσης και για την, τον απολογισμό, την ενημέρωση που μα κάνετε. Για το ΕΛΚ είναι πολύ σημαντικέ οι επιστροφέ, γιατί αν δεν μπορούν να επιστραφούν αποτελεσματικά στη χώρα καταγωγή του εκείνοι που δεν δικαιούνται διεθνού προστασία, δημιουργείται ένα μεγάλο άχθο για το συνολικό σύστημα ασύλου στην Ευρώπη. Επομένω, είναι πολύ σημαντικό να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά μα σε αυτό. Η τελευταία, μάλλον, συμφωνία υπερνησδοχή ήταν το 2014 που συνήφθη. Επομένως θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειε μα. Είναι καλό να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει συνεργασία με τι χώρες στην ανατολική γειτονία, στα ανατολικά μας σύνορα. Ωστόσο θα πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία μας με τους γείτονές μας στο νότο. Κύριε Πρόεδρε, αν δούμε και τα στοιχεία από το διάρκεια του 2019 είχαμε πάνω από 10.000 εισόδου από την Αλγερία και το Μαρόκο, που χώρες που έχουν ποσοστά 5 και 10% αντίστοιχα αναγνώρισης διεθνού προστασίας. Και είχαμε ουσιαστικά 4 στους 5 Αλγερινούς να παραμένουν στην Ευρώπη. Αν δούμε τις ε, του αριθμού των επιστροφών. Το οποίο θα σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα παραμείνουν στην Ευρώπη εξαρτήτω των διαδικασιών μα και των συμφωνιών μα. Επομένω, θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα να βελτιωθούν τα αποτελέσματα. Το ερώτημα είναι πώ. Πρέπει πρώτα απ' όλα να βελτιωθεί η οδηγία για τι επιστροφέ. Ελπίζω αυτό να το προωθήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Αλλά Επίσης υπάρχουν και άλλες δυνατότητες βελτίωσης των διμερών σχέσεων με τις χώρες αυτές. Για παράδειγμα κάτι που ποτέ δεν κατάλαβα και ελπίζω ίσως να μπορέσετε να με βοηθήσετε εσείς. Όταν έχουμε τη συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοτονού. Όλες αυτές οι χώρες είχαν συμφωνήσει ε, διαδικασίες επανεισδοχής για παράτυπα διαμένοντες ε, οι που βρίσκονται στην Ευρώπη και αντιστοιχώ η Ευρώπη από τη σειρά τη είχε συμφωνήσει. Επομένως αυτό το σκέλος της συμφωνίας Κοτονού γιατί δεν έχει εφαρμοστεί και έχουμε ξεκινήσει να διαπραγματευόμαστε ή τέλο πάντων θα ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση μέσα στο 2020 για μια νέα συμφωνία με τις χώρες αυτές. Και το ερώτημα είναι σε αυτή τη νέα συμφωνία Ποια είναι η προσέγγιση μας, πώς θα διαπραγματευτούμε με τις χώρες αυτές διατάξεις για τις επιστροφές και τις επανεισδοχές που να εφαρμόζεται στην πράξη. Δεν αρκεί να έχουμε διεθνείς συμφωνίες, πρέπει να εφαρμόζονται και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι τρίτες χώρες εναντί μας. Κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία κυρία Παρέτ. Κυρία Παρέτ. κοιτώντας τα, τους αριθμιστικά στοιχεία βέβαια, πέρα από τα αριθμητικά στοιχεία που μας ε, έδωσε ο κύριος Λέναρς, υπάρχουν και άλλες ε, περιπτώσεις τις οποίες δίνεται ανθρωπιστικό καθεστώς χωρίς και δεν προχωρούμε σε επανεισδοχή ή επιστροφή. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, όταν έχουμε τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες επανεισδοχής, πώς εισάγουμε ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. Μιλούμε για παράδειγμα να συνάψουμε ε, συμφωνίες επανεισδοχής με χώρες όπως το Μαρόκο. Μήπως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και άλλες παραμέτρους έτσι ώστε να είναι πραγματικά θελοντική αυτή η διαδικασία. Μιλάμε συχνά για το πόσο σημαντικό είναι να φτιάχνουμε ασφαλές και ε, νόμιμες διόδους και έχουμε 60.000 περιπτώσεις από το 2015 μέχρι το 2019 ανθρώπων που επαναγκαταστάθηκαν, το οποίο σημαίνει περίπου 7.000 άτομα το χρόνο, το οποίο ε, ε, ε, για ανακράτος μέλος να το δει κανείς, είναι λιγότερο από 800 άνθρωποι. Αυτή είναι η συνεισφορά της Ευρώπης στο πρόβλημα της, στο διεθνές πρόβλημα της μετανάστευσης και αν αυτό, αυτή είναι η κατάσταση είναι λυπηρό γιατί ζητούμε από άλλες χώρες των κόσμο να κάνουν πολλά περισσότερα. Επομένως θα πρέπει να φροντίσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα με το οποίο δεχόμαστε ανθρώπους. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε ε, πώς χρησιμοποιείτε το Ταμείο Άμυφ. Έχουμε κάποιες πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι οι επιστροφές στις χώρες προέλευσης, καταγωγής, προβλέπεται ένα ποσό 953 εκατομμυρίων ευρώ στην περίοδο μιας τετραετίας μέχρι το 2019. Θα ήθελα να μου πείτε για τους άλλους τομείς του τομείου ΑΜΙΦ. Ποια είναι τα κονδύλια, ποιο είναι το ύψος των κονδύλιων. Για παράδειγμα, για την ένταξη στις ευρωπαϊκές χώρες των ανθρώπων αυτών. Τι ξοδεύουμε. Και επίσης, για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν μιλούμε για επιστροφές, όταν αναφέρεται αναφερικά στοιχεία, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε. Μιλούμε μόνο για επιστροφές προς τις χώρες προέλευσης και όχι για επιστροφή από το ένα κράτος μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κράτος πρώτης άφηξης. Θα ήθελα να μου το διευκρινίσετε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πάριατ. Κυρία Πάριατ. Νομίζω, λέει κυρία Ινφελτ, νομίζω όλοι συμφωνούμε για το πόσο σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα επιστροφών που να λειτουργεί. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα εξέταση των ετοιμάτων ασύλου, εάν κάποιο δεν δικαιούται να παραμένει, θα πρέπει να πλάβνεται. Βεβαίω, το ζήτημα δεν είναι να κοιτάμε μόνο τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία. Και για αυτά έχω κάποιε ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το νομικό καθεστώς αυτών των συμφωνιών. Εάν δεν απατώμα υπάρχουν 16 επίσημες συμφωνίες, ενώ άλλες είναι διευθετήσεις με ονόματα του τύπου μια κοινή διακήρυξη για το μέλλον. Θα ήθελα να μου πείτε αυτές οι 7 ποιο είναι το νομικό τους στάτους. Μπορεί να τις εξετάσει για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή προβλέπονται άλλες δικλείδες ασφαλείας για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα έρθω επίσης και να έρθω για το ζήτημα της ε, ένταξης. Εγώ θα σας μιλήσω πιο συγκεκριμένα για το ζήτημα των, παιδιών από το Αφγανιστάν και την επιστροφή των παιδιών προς το Αφγανιστάν. Λέγεται ότι το 3 τέταρτα των παιδιών που, ε, από, τους οποίους, από τα οποία λεφθεί συνέντευξη ε, δήλωσαν ότι δεν αισθάνθηκαν ασφαλή σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές σε πολλές περιπτώσεις αυτά στάλησαν στην, στο Αφγανιστάν είτε μόνα τους είτε με αστι, αστι, συνοδεία αστυνομικών. Μόνο τρία από τα 53 παιδιά που στείλαμε πίσω στο Αφγανιστάν ε, εντάχθηκαν σε κάποιο πρόγραμμα ένταξή τους στο Αφγανιστάν. Μόνο 16 πήγαν σχολείο. Έγιναν προσπάθειες από ορισμένους να τους στρατολογήσουν για να προβούν σε πράξεις βίας και πρόκειται για παιδιά που τώρα πια λένε ότι δεν θέλουν να ξαναπροσπαθήσουν να πάνε στην Ευρώπη. Είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτό είναι βιώσιμη κατάσταση και τι είδους παρακολούθηση κάνει η Επιτροπή. Δεν φαίνεται να γίνεται πραγματική παρακολούθηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο, για το τι θα συμβεί σε αυτούς τους ανθρώπους από την στιγμή που τους επιστρέφουμε στις χώρες αυτές και σας έφερα το παράδειγμα του Αφγανιστάν ε, γιατί γνωρίζουμε την ιδιαίτερα δυσμενή θέση των γυναικών και των κοριτσιών στη χώρα αυτή. Πώς μπορούμε να έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή με, αυτές, με αυτή την κατάσταση. Αναφερθήκατε στη συνεργασία με την Τουρκία. Εν τέλει, γνωρίζουμε ότι έχουμε επενδύσει σημαντικά στις σχέσεις με την Τουρκία και στη συνεργασία μαζί της για να δέχεται ανθρώπους ε, που ε, απελάβνουμε, όμως γνωρίζουμε ότι ο αριθμός αυτών που η Τουρκία δέχεται ως επανεισδοχές παραμένει πολύ μικρός, επομένως θέτω το ερώτημα, αξίζει τελικά αυτή η συνεργασία μαζί τους. Ευχαριστώ. Κυρία Στέκ, θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ την κυρία Μπρέτ και προσβλέπω πραγματικά στη συνεργασία μαζί σας τα επόμενα χρόνια. Και φαντάζομαι ότι ήδη και η παρουσίαση εδώ ήταν ε, μια σημαντική επίδοση. Έχουμε σημαντικές ερωτήσεις βέβαια να σας κάνουμε. Ένα από τα θέματα είναι ότι η συνεργασία με τις ε, χώρες διαμετακόμισης πρέπει να έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από ότι η συνεργασία με τις ε, χώρες προέλευσης. Ενώ παλαιότερα η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστηνε στο Συμβούλιο να εστιαστεί στις χώρες προέλευσης, γιατί αφενός υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία διαπραγμάτευσης και εκεί δημιουργούνται οι κίνδυνοι για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί προφανώς ο κόσμος είναι στις χώρες του. Αυτό δεν το ακολούθησαν τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο ως Συμβουλή. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές συμφωνίες επανειστοχής με τις ε, ενδιάμεσες χώρες και τις χώρες προέλευσης και με τις δύο ως επιτοπλιστών δηλαδή. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό. Ακόμα και σε μα, συμφωνίες επανεισδοχής δεν βλέπουμε αυτή την υποχρέωση να επιστραφεί ο κόσμος στην χώρα προέλευση. Δεν σας φαίνεται ότι αυτό θα ήταν λίγο πιο λογικό. Κοιτώντα ε, και τις ε, συμφωνίες επανειστοχής βλέπουμε ότι μπορούν οι χώρες να χρησιμοποιήσουν οι επίσημες ή οι ανεπίσημες συμφωνίες. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν προωθούμε τη χρήση των επίσημων συμφωνιών αφού υπάρχουν. Και πείτε μας επίσης, οι επίσημες ε, συμφωνίες επανεισδοχής σε ποιες περιπτώσεις και πόσες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται. Πείτε μας κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τις εταιρικές σχέσεις τις οποίες αναφέρατε. Προφανώς ε, χρησιμοποιείται οποιαδήποτε επιρροή και συζητήσαμε με τον Τζόνσον τα θέματα αξιολόγηση κινδύνου, γιατί αυτές οι συμφωνίε έχουν ε, το αποτέλεσμα να παραμένουν οι άνθρωποι παγιδευμένοι σε κάποιες χώρε διέλευση, χωρί πρόσβαση στο άσυλο. Προτίθεστε λοιπόν να κάνετε μια αξιολόγηση κινδύνου προτού ξεκινούν αυτές τις συνεργασίες και να παρακολουθούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο για τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την επίτευξη τη συμφωνία αυτή. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ανεξαρτησία. Δύο σύντομα στοιχεία τώρα. Θα ήθελα να τονίσω αυτά που είπε η κυρία Ιντφέλτ. Έχω και εγώ την ίδια ερώτηση να κάνω. Για τα παιδιά επιτέλου, νομίζω ότι είναι πολύ ανησυχητικό το θέμα αυτό. Και στην οδηγία για τι επιστροφέ αναφέρεται ότι προφανώ θα πρέπει να επικρατεί ω πρώτη στην προτεραιότητα το συμφέρον του παιδιού. Αυτό Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο θα το κοιτάξετε στην επόμενη συνάντηση. Και ένα θέμα σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σε ό,τι αφορά την τουρκική κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και α, Τουρκίας. Έχουμε λάβει τις ειδήσει ότι η Μέρκλ σχέθηκε στον Ερντογάν και οικονομικές δυνατότητες για την δημιουργία κέντρων υποδοχής στην Βορειοανατολική Συρία. Θα μας ε, πείτε, μπορείτε να μας εξασφαλίσετε ότι δεν θα δαπανηθούν πόροι εκεί στη Συρία από την τουρκική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος. Συνάδελφοι, ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να διακόπτω. Αλλά να έχετε υπόψη ότι είναι πολύ βαρημένη η ημερήσια διάταξη σήμερα. Συζητάμε λοιπόν ε, αυτά τα καταπίδωτα θέματα, την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι συμφωνίες επανεισδοχής και επιστροφής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά είναι παράλληλα με τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει τα κράτη-μέλη. Αλλά να έχετε υπόψη ότι θα πρέπει να γίνει και κάποια συζήτηση και για το σημείο 8 για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας. Έχουμε ήδη την παρουσίαση του Πέταρ Βιντενοφ, ο οποίος είναι ο εισηγητής για το θέμα αυτό. Και το 9. Παρουσίαση της ε, συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκορωσίας και τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων. Επίσης και εδώ η κυρία Παριάτ θα μας παρουσιάσει τι συμβαίνει. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Και μετά τους συντονιστές παρακαλώ, όσοι θέλουν να κάνουν ε, ρωτήσεις παρακαλώ να το κάνουν εν συντομία. Γιατί έχουμε και το θέμα της κυρίας Σίπελ μετά. για τα e-evidence, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικέ υποθέσεις. Μετά έχουμε και τις ηλεκτρονικέ ψηφοφορίε μετά την παρουσίαση του κ. Γκόσταϊλ από την Europol και όλα αυτά πριν από τις 11.30. Σας παρακαλώ. Δεν μπορείτε να μιλάτε τρία λεπτά ο καθένα. Θα πρέπει τώρα να ακούσουμε τον επόμενο κύριο συνάδελφο, τον κύριο Βέστ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πάριατ, που ήρθατε εδώ σήμερα. Να σα ε, πω ένα πράγμα, κύριε Λόμπο Αγγιλάρα. Αν δεν κάνετε τόσες πολλές εξηγήσει για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρόνο, θα μπορούσαμε να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Μπορούμε να τη διαβάσουμε και μόνοι μας την ατζέντα. Δεν χρειάζεται να να κάνετε τόσο μεγάλες εισαγωγές. Μπορείτε να είστε πιο σύντομο στο συντονισμό της συζήτηση. Δεν χρειάζεται να μου πείτε εσεί τι είναι δημαγωγία και τι δεν είναι. Και όταν μας λέτε ότι η κρίση η μεταναστευτική ήταν στο ύψιστο σημείο το 2015 και ότι απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ψέμα. Γιατί άνοιξε λοιπόν τα σύνορα η κυρία Μέρκελ, γιατί έγιναν όλα αυτά που έγιναν στην Ουγγαρία, γιατί είχαμε ε, ε τρομοκράτες στην Γερμανία με 27 διαφορετικές εθνικότητες. Αυτό καταδεικνύει ότι έχουν αποτύχει πλήρως τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, ελέγξουν την κατάσταση το 2015-2016 και η συμφωνία με την Τουρκία. Αυτό, ακριβώ καταδεικνύουν. Κυρία Παριάτη, μια σύντομη ερώτηση έχω να σα κάνω. Έχουν γίνει ερευνέ για το... για τους νόμιμους μετανάστες οι οποίοι ε, εντάχθηκαν ε, στο ε, πρόγραμμα επαναγκατάστασης. Είπατε ότι είναι 75.000 άτομα από το 2015. Ε, είναι ακόμα στις χώρες που υποτίθεται ότι ήταν μετά την επαναγκατάσταση ή έχουν ε, μεταναστεύσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα μπορούσατε να μας δώσετε τα στοιχεία σχετικά για το ποιες χώρες έχουν τελικά υποδεχτεί πόσους ανθρώπους στα πλαίσια του προγράμματος επανεγκατάστασης. E Εκπρόσωπη του ECR, η κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διευθυντρία, για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Το ECR υποστηρίζει την ε, επιστροφή επιστροφών, την πολιτική επιστροφών για την επιστροφή των ε, παράνομων μεταναστών στις χώρες τους. Ε, και είμαστε υπέρ της αναθεώρησης της οδηγίας για τις επιστροφές επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Μα, λίγα και καλά, λέει ο πρόεδρος. Η Γκουε, η κυρία Πιόρκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω καταρχάς για τα, για τα στοιχεία που λάβαμε, για τα έγγραφα που λάβαμε, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και να αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία ανέφεραν οι συνάδελφοι. Καταρχάς να πω ότι πιστεύω ότι σε κάποιες περιπτώσεις όταν ακούμε για τις επιστροφές θα ήθελα ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ήταν τουλάχιστον κατά το τόσο αποτελεσματικά για την αξιοπρεπή υποδοχή των ανθρώπων αυτών. Δεν θα είμαστε εκεί που είμαστε σήμερα αν το πετυχαίναμε αυτό. Και κάποιοι θέλουν να κάνουν μια σύνδεση μεταξύ της νομιμότητας του συστήματος ασύλου και του επίπεδου επιστροφών. Δεν έχουμε όμως οποιοδήποτε στοιχείο που το υποστηρίζει αυτό. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε ξενοφοβία και ο, ο άνθρωπος χάνει την ανθρώπινη διάστασή του. Αυτό είναι το πρόβλημα στο σύστημα ασύλου μας. Δύο θέματα ήθελα να θίξω. Κάποια τα είπαν και οι συνάδελφοι και η συγκεκριμένα η κυρία Ιντφέλτ σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν και την επιστροφή παιδιών. Και είναι σαφέ ότι πολλοί από αυτού από εμά που έχουν διαβάσει αυτή την ε, έκθεση, έχουμε δει παραδείγματα και υποθέσει που καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι το Αφγανιστάν δεν είναι μέρο να επιστρέφονται τα παιδιά. Αυτό είναι το συμπέρασμα, όπω και αν το δούμε από τη χώρα μου, τη Σουηδία, να σας πω ότι το θέμα αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ε, παίρνουμε τα παιδιά, τα βγάζουμε από το σχολείο, τα βγάζουμε από την οικογένειά τους, την καινούργια οικογένειά τους, από τον περίγυρό τους και τα στέλνουμε στο Αφγανιστάν ε, σε τελείως μη ασφαλείς συνθήκες και πραγματικά είναι τεράστιες οι διαμαρτυρίες. Ελπίζω να σταματηθούν, να σταματήσουν αυτά σύντομα. Και ελπίζω πραγματικά να μην χωράει καμία αμφιβολία αυτό σε ό,τι αφορά τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκίας. Δεδομένου των περιορισμένων αριθμών επιστροφών, αξίζουν τον κόπο τα χρήματα που τα πανούμε. Δεν ε, είμαι κατά, αλλά η νομιμότητα που δώσαμε και η ισχύ που δώσαμε στον Ερντογάν στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής αξίζουν τον κόπο. Θεωρώ ότι η απάντηση είναι ένα σαφές και χειρό όχι Κυρία Μπιόρκ, βλέπω ότι το λόγο ζητάει άλλος ένας συνάδελφος. Εν συντομία, ωστόσο, γιατί έχουμε και τον κύριο να έχετε μετά το λόγο. Θέλετε να αναβραθείτε στο θέμα αυτό. Μάλιστα. Ναι, και εσείς για το θέμα αυτό. Μάλιστα. Πρώτο πάρτε το λόγο για τη Λευκορωσία. Άρα, ο κύριος Τουντεράτσο και μετά ο κύριος Βιτανινό. Αλλά μετά έχουμε και τη Λευκορωσία και τις θεωρήσεις. Ο κ. Βουτάνοφ είναι υπεύθυνο για την ε, Λευκορωσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Εδώ έχω πολύ συγκεκριμένε απόψεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Παριάτη για την ενημέρωση και ήθελα να μου πείτε περισσότερα για το σύμφωνο. Είπατε ότι η επανεισδοχή θα είναι μέρος του νέου συμφώνου. Το είπα και προηγουμένως, εάν στο σύμφωνο αυτό η επανεισδοχή και οι επιστροφές δεν είναι σωστά εξισορροπημένες ε, με τα υπόλοιπα του ασύλου και δεν πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες, τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα που στις πρωτεύουσε ζητούν για το σύμφωνο, θα πρέπει να περάσουν σε διεξοδικές συζητήσεις για τα θέματα τη μετανάστευση και τι είναι ε, διατεθειμένοι να διαθέσουν, να προσφέρουν για το θέμα αυτό. Διότι χωρί σύμφωνο η επιτυχία που θέλουμε με τι τρίτε χώρε δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πραγματικότητα. Ευχαριστούμε κύριε Τοντοράτσι. Βίτανοφ, ευχαριστώ πολύ γρήγορα ένα σχόλιο και τη ρωτήσεις. Είπατε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για, την, για τις απεινές δοχές. Οι Τούρκοι είπαν ότι δεν θα ε, εφαρμόσουν τις διατάξεις για την επανεισδοχή αν δεν έχουν απελευθέρωση των θεωρήσεων. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα λοιπόν για τη διαδικασία απελευθέρωσης των θεωρήσεων με την Τουρκία και για τον τροποποιημένο κώδικα για τις θεωρήσεις, των θεωρήσεων που θα θέσετε σε εφαρμογή την επόμενη εβδομάδα και προβλέπει ένα νέο σύστημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέτε ότι εκεί θα μπορούμε να πιέσουμε για τις περιπτώσεις επανεισδοχής. Τι θα γίνει εκεί με την Τουρκία και τη διαδικασία επελευθέρωσης των θεωρήσεων. Και η δεύτερη ερώτηση είναι για τη μελλοντική συμφωνία. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκο. Σκοπεύετε να ξεκινήσετε και πάλι διαπραγματεύσεις. Από τι εξαρτάται αυτό. Και ένα γενικό σχόλιο Νομίζω το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, συμμετέχει ενεργά και να ενημερώνεται για τι εξελίξει των δημοτεύσεων ατύπων και επισήμων συμφωνίων επανεισδοχή και συμφωνώ εδώ με την κυρία Στρίκ, διότι όποτε ε, είναι αυτό δυνατό θα πρέπει να υπάρχουν επίσημε συμφωνίε παρά το να έχουμε άτυπε διευθυντήσεις και διαδικασίε για να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλου του κόσμου. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου. Δεν βλέπω άλλοι να σηκώνουν το χέρι. Κυρία Παριάτ, προτείνω το εξή. Έχετε μόλις ξεκινήσει και μάλιστα δύσκολα γιατί πήρατε μια σειρά από σχόλια και πολύ συγκεκριμένες, πάρα πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα έλεγα να λάβετε τώρα το λόγο για να τις απαντήσετε και μετά να σας ξαναδώσουμε το λόγο για να μπορέσετε να μιλήσετε και για την περίπτωση της Λευκορωσίας και για την περίπτωση απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Με αυτή τη σειρά θα μπορέσουμε να ακούσουμε αναλόγω και του εισηγητέ μα. Τον κύριο Βέτανοφ για τι θεωρήσει για τη Λευκορωσία και τον κύριο Χουκ για το θέμα τη διευκόλυνση των θεωρήσεων. Συμφωνείτε? Ωραία. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ όλου για τι ερωτήσει σα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ή δυνατόν όλε και θα αφήσω και τον συνάδελφο να σα δώσει κάποιε τεχνικέ ε, διευκρινήσει για την ε, συνεργασία με τους γειτονές μας, Μαρόκο και Αλγερία, κύριε Λέναρτ, ε, υπόθηκε και σε άλλη ερώτηση για τη συμφωνία με την Αλγερία. Ναι, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, ιδίω με το Μαρόκο. Αυτό όμως είναι ένα συνολικότερο σχόλιο που θέλω να κάνω. Πρέπει να έχουμε μια σφαιρικότερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες και να συμπεριλαμβάνουμε όχι μόνο τα θέματα μετανάστευση στην όλη συζήτηση, αλλά συνολικότερα να κοιτάξουμε πώς συνεργαζόμαστε μαζί τους. Οι συζητήσεις με το Μαρόκο, όπως ξέρετε, είχαν μπλοκαριστεί επί σειρά ετών. Τώρα μπορούμε να ξαναρχίσουμε και να δούμε και μια σφαιρικότερη συμφωνία εταιρική σχέση. Η συζήτηση για τα θέματα τη μετανάστευση μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο. Και έτσι θα αναζητήσουμε μια εξισορροπημένη μορφή συνεργασία μαζί του. Αυτή την προσέγγιση θέλουμε να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Αναφέρατε τη Συμφωνία Κοτονού Εγώ θα ήθελα να το ε, θέσω λίγο ευρύτερα. Όλα τα κράτη έχουν κυρώσει τη Συμφωνία της ε, Γενέβης. Όλοι είναι συμβαλόμενα μέρη. Αυτή είναι η νομική βάση. Αυτή είναι η κατάλληλη νομική βάση για να βεβαιωθούμε ότι κόσμος που δεν έχει δικαίωμα να παραμείνει σε άλλη χώρα ε, απομακρύνεται. Βασιζόμαστε στο διεθνές δίκαιο. Βάσει του διεθνούς δικαίου ε, Περιμένουμε όλες οι χώρες να σεβαστούν αυτή τη συμφωνία. Και για τις ερωτήσεις διμερών συμφωνιών, επανεισδοχής ή σχετικών διευθετήσεων, οι συμφωνίες αυτές, οι διευθετήσεις, σκοπό δεν έχουν να επιλύσουν τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με τις περιπτώσεις αυτές στέλνουμε πίσω κόσμο που ε, η περίπτωσή τους έχει εξεταστεί ενδελεχώς σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα ασύλου που έχουν. Με όλους τους απαραίτητους ελέγχους που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Υπήρξαν ε, συμφωνίες που σκοπό είχαν να κοιτάξουν τις διαδικασίες των επιστροφών και σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχει ακόμα μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να γίνουν και πρέπει να επαληθευτούν ε, περαιτέρω. Όμω ε, τον κόσμο αυτόν τον επιστρέφουμε με τρόπο αξιοπρεπή. Σε αυτό σας καθησυχάζω. Ισχύει για όλες μας τις συμφωνίες. Και ή δυνατόν θέλουμε συμφωνίες που να καλύπτουν τα πάντα. Εκεί ζητούμε τη σύμφωνη γνώμη σα και αυτή είναι σίγουρα η εναλλακτική που προτιμούμε. Όμως δεν είναι πάντοτε εφικτό και όταν δεν είναι εφικτό, όταν μια τρίτη χώρα δεν θέλει να συνάψει συμφωνία, τουλάχιστον καλό είναι να έχουμε κάποια διευθέτηση, η οποία είναι ένα εργαλείο μη δεσμευτικό, είναι διοικητικού τύπου. Επιτρέπει τουλάχιστον να θέσουμε κάποιες προϋποθέσεις για το πώς διοργανώνεται η επιστροφή και κοιτάζουμε αν μπορούμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες για την επιστροφή των προσώπων στις διάφορες χώρες ή να οργανώσουμε τις επιστροφές με βάση κάποια κριτήρια, διοικητικά και τεχνικά. για το Ταμείο ΑΜΕΦ. Εγώ το βρίσκω κάπω αρκετά καλά εξισορροπημένο, αλλά θα αφήσω τον συνάδελφο να σας πει περισσότερα γι' αυτό. Εάν καλά θυμάμαι, έχουμε χρηματοδότηση 943 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το κλασικό ποσό, αλλά έχουμε πολύ μεγαλύτερα ποσά από την αλληλεγγύη για την επανατοποθέτηση και ε, τα θέματα επιστροφής, 5 εκατομμύρια ευρώ. Ε, νομίζω ότι είναι αρκετά καλή η ισορροπία που έχουμε πετύχει. για τις προϋποθέσεις επιστροφών προς τις χώρες και οι συμφωνίες αυτές σκοπό είχα να υπογραφούν κατά προτεραιότητα με τις χώρες προέλευσης και όχι με χώρες διέλευσης, με μόνο εξαίρεση την Τουρκία. Οι συμφορίε αυτές με τις χώρες προέλευσης είναι ο καλύτερος τρόπος να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος επιστρέφεται σε ε, μια χώρα που του είναι εκεί, που την ξέρει καλά και όχι σε μια χώρα την οποία απλώ πέρασε και έκανε μια διέλευση. Αφγανιστάν. Η προηγούμενη δουλειά μου ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια. Γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Και πάλι εδώ έχουμε νομοθεσία που ισχύει και πράγματι όταν κάποιος δεν έχει δικαίωμα νόμιμες παραμόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να επιστρέψει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και είναι και όλο σκοπός αυτών των συμφωνιών και των διευθετήσεων είναι όσο μπορούμε να συνοδεύσουμε τον άνθρωπο αυτό. Ακόμα και οικονομική υποστήριξη δίνουμε. Τον κόσμο που επιστρέφουμε στις διάφορες χώρες, κοιτάμε να τον βοηθήσουμε. τους προσφέρουμε κάποιες ε, συνθήκες διαβίωσης στις χώρες τους. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η κατάσταση στο Αφγανιστάν σίγουρα δεν είναι ικανοποιητική. Απέχει πολύ. Ε, προσπαθούμε με τους συναδέλφους από άλλες υπηρεσίες όπω την προηγούμενη Γενική μου Διεύθυνση και την υποστήριξη που προσφέραμε στα πλαίσια τη αναπτυξιακή πολιτική, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, αντιμετωπιστούν ζητήματα μακροπρόθεσμης ανάπτυξη. να μπορεί ο κόσμος να έχει κάποια ανθρωπιστική υποστήριξη. Και προσπαθούμε και να έχουμε και κάποια τέτοια αναπτυξιακή πολιτική, ώστε οι λύσει μακροπρόθεσμα να είναι βιωσιμότερε. Δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε όλα για μια, μια συμφωνία πανεισδοχή. Είναι σαφέ ότι οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από τις χώρες τους διότι δεν μπορούν εκεί να κερδίσουν τα προστοζήν. Και γι' αυτό έχουμε τις συμφωνίες επανεισδοχής για να προσπαθήσουν ε, να, να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε μια καλύτερη ευκαιρία στη χώρα προέλευσης. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε δεσμευτεί να παρακολουθούμε στενά το πώς εφαρμόζονται οι συμφωνίες στις χώρες προέλευσης και θα συνεχίσουμε να το εξετάζουμε το θέμα αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την Τουρκία, αν αξίζει τον κόπο Νομίζω εδώ πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο ευρύτερα. Η υποστήριξη που έχουμε προσφέρει στην Τουρκία επιτρέπει να υποστηριχθεί 1,7 εκατομμύρια κόσμος οι οποίοι παραμένουν στην Τουρκία. Η Τουρκία έχει υποδεχτεί 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Οι άνθρωποι αυτοί, χάρη στην υποστήριξή μας, μπορούν να έχουν κάπως καλύτερη μεταχείριση και να υποφεληθούν από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ώστε να παραμείνουν στην Τουρκία όσο η κατάσταση στην Συρία δεν βελτιώνεται. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τα πράγματα λιγάκι σφαιρικότερα. Ε, Ποιο είναι ο αντίκτυπο, α πούμε, τη ε, διευκόλυνση Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Τώρα για τα κονδύλια και το κατά πόσον θα χτίσουμε εγκαταστάσει υποδοχή στα βορειοανατολικά τη Συρία. Στην Τουρκία θα δαπανηθούν τα χρήματα, όχι στη βορειοανατολική Συρία. Δεν θα υπάρξει εκεί επανοικοδόμηση. Δεν θα δώσουμε τίποτα για ανοικοδόμηση της χώρας ε, στα, στα βορειοανατολικά της Συρίας. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. για το πόσο κόσμο έχουμε επιστρέψει. Δεν ξέρω αν έχουμε σύστημα παρακολούθησης γι' αυτό. Είναι αρκετά περίπλοκο να υπολογίσουμε, αλλά ευχαρίστω να το συζητήσω διμερώ με όποιον από σα θέλει, για να δούμε τι λεπτομέρειε και πώ ακριβώ εφαρμόζονται τα πράγματα. Και για το σύμφορο της μετανάστευση Όπως προείπα, το σύμφωνο της μετανάστευσης το μελετάμε ήδη. Η προσέγγιση που θέλουμε να ακολουθήσουμε είναι σφαιρική, είναι συνολική. Συμφωνώ με όλους σας ότι προκειμένου να έχουμε ομαλότερη επιστροφή όσων δεν έχουν δικαι... νόμιμο δικαίωμα παραμονής ε, στην επικρατειά μας πρέπει να ασχοληθούμε με τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης, ε, με την, ε, με την κατάσταση, με την επανεισδοχή, με άλλους τρόπους ανθρωπιστικής ε, με, κατάστασης του κόσμου. Θα κοιτάξουμε τι διαδικασίες μπορούμε να συμπεριλάβουμε στο σύμφωνο. Και τέλος, Από την πλευρά μου επιβεβαιώνω ότι πολύ συστηματικά θα σας ενημερώνουμε και θα φροντίζουμε να γνωρίζετε τα των διαπραγματεύσεων στο μέλλον. Προς στιγμήν δεν υπάρχουν πολλές εξελίξει. Ο σκοπός μας πάντως είναι να συνεχίσουμε και ελπίζουμε όλες οι χώρες να έχουν διάθεση συνεργασία. Ο στόχο είναι να δημιουργηθεί μια σφαιρικότερη προσέγγιση και με άλλα εργαλεία για να διευκολύνουμε τα πράγματα. Και να δώσω το λόγο και στον ε, Ευχαριστούμε κυρία Παριάτ. Ε, πραγματικά έχουμε καθυστερήσει. Αν μπορείτε λίγο να επιταχύνετε, διότι υπάρχουν δύο ακόμα σημεία προ εξέταση στην υπηρεσία διάταξη. Κυρία Παριάτ, θα πρέπει να δούμε τη συμφωνία με τη Λευκορωσία και την έκδοση των θεωρήσεων. Έχουμε εδώ τους εισηγητέ μας. Ε, θα υπάρξουν εκεί και ερωταπαντήσει και τα μέλη έχουν δικαίωμα να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν πολύ γρήγορα. Δύο λεφτά μόνο για τρεις ερωτήσεις. Το είπε η κυρία Παριάτ. Το Ταμείο Επανένταξης με τη Μετανάστευση 900 εκατομμύρια ευρώ είναι απόλυτα ε, λογικό, 943 μάλλον, τα περισσότερα πηγαίνουν για την επανεγκατάσταση και για την επανένταξη. Είναι λογικό το ποσό και μετά τη συνάντηση μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για τον κύριο Βετανόφ και για τις ερωτήσεις του για την Τουρκία. Ξέρετε ότι η απελευθέρωση είχε να κάνει με κάποιους δείκτες συγκριτική αξιολόγησης, τους κοιτάμε ακόμα, δεν υπάρχει περισσότερη πρόοδος συνολικά. Ε, κοιτάζουμε τη διαδικασία απελευθέρωσης θεωρήσεων με την Τουρκία. Το άρθρο 25α του τροποποιημένου κώδικα θεωρήσεων επιτρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στην έκδοση θεωρήσεων εφόσον χρειαστεί για να ασκηθεί πίεση σε τρίτες χώρες, να ε, εφαρμόζουν διαδικασίε επανειστοχή, επιστροφέ και επανειστοχέ, όμω αυτό πρέπει να λάβει υπόψη συνολικά πώ είναι η σχέση μα με μια δεδομένη τρίτη χώρα. Και βεβαίω, ε, υπό αυτή την οπτική γωνία, θα δούμε συνολικά τη σχέση μα με την Τουρκία για την περίπτωση των ε, θεωρήσεων και αν θα υπάρξουν διευκολύνσει ή περιορισμοί. Τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 20 δευτερόλεπτα, 25 δευτερόλεπτα. Όπω γνωρίζετε πολύ καλά, και το εξηγήσε και η Μονίκ, οι συμφωνίε επανεισδοχή δεν είναι το εργαλείο για να επιβάλλουμε το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν ληφθεί απόφαση επιστροφή και στη διαδικασία ασύλου και επιστροφή, τα δικαιώματα των μεταναστών πρέπει να γίνονται σεβαστά. Τα λαμβάνουν υπόψη του στα δικαστήρια και οι εθνικέ διοικητικέ αρχέ. Φυσικά όλε οι δυνατότητε για τι μετέπειτα υποβολέ αιτήσεων ή για έφεση κατά τη απόφαση ε, προβλέπονται. Πάντω, μια από τι προτεραιότητε για το μέλλον είναι να βελτιώσουμε την υποστήριξη προ την επανεισδοχή, την επανένταξη και τα προγράμματα οικειοθελού επιστροφής. Θα κοιτάζουμε λοιπόν ε, τι γίνεται με τα παιδιά και τους ανθρώπους που επιστρέφουν σε τρίτες χώρες. Εκεί πρέπει να παρακολουθούμε στενά το τι συμβαίνει και να φροντίζουμε σε ποιο πλαίσιο εντάσσονται. Ε, εκεί πρέπει να κοιτάζουμε την πολιτική επανένταξή μας. Ευχαριστούμε και τους δύο εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Ιστορικών Υποθέσεων. Εσάς, κυρία Παριάτ. Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα που έχουμε μπροστά μας, ε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα. κυρία Παριάτ, θα μας παρουσιάσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα τη Συμφωνία Πανεσδοχής Λευκορωσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, μετά θα ακούσουμε τους συζητητές μας. Έχετε το λόγο και πάλι αλλά γρήγορα. Συνοπτικά, όχι όλα. Λοιπόν, σύντομα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε μια διαπραγμάτευση, είχαμε μια διαπραγμάτευση πάνω από πέντε χρόνια με τη Λευκορωσία και για την διευκόλυνση θεωρήσεων και για την Συμφωνία Πανεισδοχής. Χωρίς να μακρηγορούμε όμως, Ολοκληρώθηκαν αυτές οι διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο του 2019 και καταλήξαμε στις ε, συμφωνίες αυτές, οι οποίες είναι το ε, παύγασμα όλων των προσπαθειών που κάναμε για να φροντίσουμε να έχουμε μια καλή ε, συνεργασία με τη Λευκορωσία που είναι και η τελευταία χώρα της Ανατολικής Γειτονίας για την οποία δεν είχαμε ακόμα μια συμφωνία για τη διευκόλυνση θεωρήσεων και τις επανεισδοχές είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστηματική αυτές οι δύο συμφωνίες, δηλαδή οι επανεισδοχές και η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων να πηγαίνουν μαζί, χέρι-χέρι. Όσον αφορά τις επανεισδοχές, τα στατιστικά μας δείχνουν ότι έχουμε ήδη μια καλή συνεργασία μεταξύ Λευκορωσίας και κρατών μελών της Ένωσης, επομένως η νέα αυτή συμφωνία μεταξύ Ένωσης και ε, Δημοκρατίας της Λευκορωσίας συμπεριλαμβάνει κάποια συνήθη στοιχεία τα οποία βρίσκουμε και σε άλλες συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Όσον αφορά τη διεθνή υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και σε πρώην υπήκοους οι οποίοι έχουν απολέσει ή είχαν αποποιηθεί της υπηκότητάς τους στα μέλη της οικογένειας ανεξαρτήτως της ε, υπηκότητας και επίσης σε υπηκός τρίτης χώρας και απάτριδες ε, σε μια χρονική περίοδο μεταβατική δύο ετών. Ε, περιγράφονται διαδικασίες για την ταυτοποίηση μεταναστών χωρίς χαρτιά και ε, ασυνόδευτων ανηλίκων. Επίσης υπάρχει μια επιταχυμένη διαδικασία ε, όταν, ε, ε, για την επανεισδοχή προσώπων στα χερσαία σύνορα μεταξύ κρατών μελών και Λευκορωσίας. Θα μπορούν να χρησιμοποιούν από εκεί και πέρα το ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό, ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο εάν δεν έχει εκδώσει η Λευκορωσία ταξιδιωτικό έγγραφο εντός μιας προθεσμίας. Υπάρχει επίσης μια διαδικασία για το transit. Δημιουργείται επίσης και μια μικρή επιτροπή παρακολούθησης της συμφωνίας. Όσον αφορά τώρα την απελευθέρωση των, τους ε, καθεστώτους θεωρήσεων, προφανώς στόχος είναι να διευκολύνουμε την έκδοση ε, θεώρησης για βραχυχρόνια παρανομή ε, στη Λευκορωσία πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστρόφως οι Λευκορώσοι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται μέχρι και 30 ημέρες ε, άνευ βίζα στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Καλύπτει αυτό μια σειρά κατηγοριών ετούντων και μια σειρά ε, στόχων, ε, ε, μάλλον σκοπών επίσκεψης, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρηματίες κτλ. Μειώνεται το τέλος σε 32 ευρώ είναι μικρότερη η χρονική, το χρονικό περιθώριο που δίνεται στα προξενία για να λαμβάνουν την απόφαση, περίπου 10 μέρες. Δίνεται επίσης η δυνατότητα η χρήση, χρήσης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων με μεγαλύτερο χρονοδιάρκειας. Απλοποιούνται τα ε, έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσει κανείς για το σκοπό της ε, ε επίσκεψης για μια σειρά ε, και επίσης εξαιρούνται εκείνοι που είναι κάτοχοι ε, διαβατηρίων διπλωματικών με βιομετρικά δεδομένα. Μετά την έγκριση που, αναμένουμε να δοθεί, που δόθηκε μάλλον στις 4 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο, υπεγράφησαν από τον Επίτροπο Ιόχανσεν τα οι συμφωνίες και τον Πρωθυπουργό το ε, τη ε, της ε, Κροατίας και τον Πρωθυπουργό της Λευκορωσίας στις Βρυξέλλες. Καλωσορίζουμε την έκθεση του εισηγητή σας και ευελπιστώ ότι σύντομα θα ολοκληρωθούν και οι διαδικασίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να τεθούν σε ισχύ αυτέ οι δύο συμφωνίε όσο το δυνατόν συντομότερα. Σα ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο για αυτή την ε, γρήγορη παρουσίαση, κυρία Παριάτ. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον εισηγητή και στους κοιόδες εισηγητές. Παρακαλώ, ε, γρήγορες παρουσιάσεις με αυτή τη σειρά. Ο κύριος Βίτανοφ που είναι εισηγητής μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα, θα μακρηγορήσω και θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω όλα αυτά που ακούστηκαν. Άρα δεν θα περιγράψω το περιεχόμενο της συμφωνίας, θα ακούσαμε αυτά. Θέλω να σταθώ στα εξή όμω, Όπως αναφέρατε, είναι η μόνη χώρα της Ανατολικής γειτονία, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμφωνία επανεισδοχή. Αυτή η συμφωνία η οποία επεγράφει πριν από δύο εβδομάδες θα είναι η πρώτη τέτοια επίσημη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Λευκορωσίας για οποιοδήποτε θέμα και αν δεν απατώμε έχουμε μια συμφωνία συνεργασίας από το 1995 αλλά εξαιτία της έλλειψης συνεργασίας και έλλειψης δέσμευσης στην δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα της Λευκορωσίας είχε ουσιαστικά πάυσει η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας συνεργασίας του 1995 με μορές από την Ένωση. Καλωσορίζουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία. Πιστεύουμε πραγματικά ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη και στενότερη συνεργασία με τις ε, χώρες της Ανατολικής Γειτονίας εξαιτία ακριβώς των προ προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτέ. Εάν δεν τίνουμε μια χείρα ε, ε, συνεργασία εμεί οι Ευρωπαίοι, κάποιο άλλο θα το κάνει. Ε, Βεβαίω δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να επισημαίνουμε τι ανησυχίε μα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να είναι στοιχείο κλειδί τη μελλοντική μα σχέση με τη Λευκορωσία. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή. Με ποιον τρόπο το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ετέθη στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, δεδομένου ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας που συνεχίζει να διατηρεί τη θανατική ποινή. Όσον αφορά τώρα τη δημιουργία αυτής της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της συμφωνίας, λέγεται ότι θα αποτελείται αποκλειστικά από εκπρόσωπο της Επιτροπής με την ε, επικορούμενο από εκπροσώπους των κρατών μελών. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρχει συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες αυτές. Η ανταλλαγή απόψεων με, με την εκπρόσωπο της Επιτροπής είναι ένα καλό τρόπος να ξεκινήσει αυτή η παρακολούθηση, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε και στις μελλοντικές συμφωνίες επανεσδοχής και θεωρήσεων να υπάρχει εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο τώρα και στους Σκιώδης, μιας και οι δύο εκθέσεις αυτές είναι πολύ ε, συναφείς. Θα δώσω το λόγο στον κύριο... Στον κύριο Χουκ για την, ε, για την έκθεση για τις ε, θεωρήσεις. Σα ευχαριστώ πολύ και είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι πολλά μπορεί να κάνει ακόμα η για τη βελτίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, εξετάσουμε την πρόοδο που έχει γίνει, γιατί αυτό σημαίνει πιο στενού ε, συνδέσμου μεταξύ τη κοινωνία των πολιτών και θα ενθαρρύνει τι εξέλιξει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόεδρε, να πω ότι ε, ο κύριος Κόλοκ μας βοήθησε, ο εμπειρογνωμονάς μου στο θέμα αυτό, στο φάκελο αυτό ο οποίο φάκελο ε, παρεμπιπτόντως όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σήμαινε μεγάλε διαπραγματεύσεις. Ξεκίνησε το 2010 να συζητιέται, 2014 ε, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, πάνω από πέντε χρόνια. Έχουμε ένα επεξηγηματικό σημείωμα τη ε, κυρίας Κώστα από τη Γραμματεία. Και τα βασικά στοιχεία να αναφέρουμε ότι περιλαμβάνουν 10 μέρες για την αίτηση, μια γρήγορη δηλαδή διαδικασία, 35 ευρώ τέλος καταβολής με εξαίρεση για τα παιδιά και άλλες ευαίσθητες ομάδες και είναι πολύ πιο απλοποιημένες οι διαδικασίες. Αλλά να πούμε ότι οι θεωρήσεις δεν θα χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθεαυτή, αλλά από τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν ένα κοινό πλαίσιο για τα κράτη-μέλη. Και φυσικά η όλη διαδικασία είναι υπό αναστολή σε περίπτωση που θα ανακύψουν θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά όπως σας είπαμε το θέμα μας είναι να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθήκαν οι σκιώδες συζητητές και χαίρομαι που έξι από τις επτά πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου είπαν ότι θα υποστηρίξουν την έκθεση αυτή. Θα ψηφιστεί το Μάρτιο στην Επιτροπή ο φάκελος αυτός και μετά στην Ολομέλεια. Εγώ πολύ λυπάμαι που δεν θα είμαι πλέον παρόν λόγω του Brexit. Θα τα παρακολουθώ όλα από την τηλεόραση και ελπίζω να περάσει ο φάκελος αυτός και ήταν μεγάλη τιμή μας να εργαστούμε επί του θέματος αυτού και να είμαστε ναι, μέλος της Επιτροπής αυτής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χουκ, λέει ο πρόεδρος της Κιώδης τώρα να μας παρουσιάσουν την απόψη τους για τα δύο αυτά θέματα. Από το ΕΛΚ ο κύριος Μπλάγκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και μιλώ εξ ονόματος του κυρίου Μπλάγκα. Όχι, είστε ο κύριος Μπόγκταν, σωστά. Έχετε και τις δύο κάρτες μπροστά σας και δεν ε, καταλάβαινα ποιος ε, ακριβώς είστε. Ο κύριος Μπόγκδαν λοιπόν θα πάρει το λόγο. Θα συνεχίσω στα ρουμάνικα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βίτσενοφ για την έκθεση του Το ΕΛΚ υποστηρίζει τη συμφωνία μεταξύ Λευκορωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση για την επανεισδοχή ατόμων τα οποία διαμένουν παρανόμω. Και ο αριθμό των ε, επιστροφών που ζητείται από τα κράτη-μέλη από τη Λευκορωσία καταδεικνύουν θετικέ τάσει παρά την απουσία συμφωνίας επανεισδοχής. 89% έχει ολοκληρωθεί ε, και αναμένεται ότι το ποσοστό θα αυξηθεί αυτό μετά την Συμφωνία Πανεισδοχή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Χου και την παρουσίασή του επίση και να πούμε ότι το ΕΛΚ συμφωνεί με το προτινόμενο κείμενο τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λευκορωσίας για την ευκολύνση στι θεωρήσει. Αν δούμε το ποσοστό άρνηση ε, θεωρήσεων για του πολίτε τη ε, Λευκορωσία το 2018, μιλάμε μόνο για πολύ πιο μικρά ποσοστά σε σχέση με το 9,8 που ήταν στο παρελθόν. Καταλαβαίνουμε την κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λευκορωσία, αλλά να μην ξεχνάμε ότι και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στη δεκαετία του 90 αντιμετώπιζαν παρόμοια θέματα. Και σήμερα πρέπει να πούμε ότι είναι πλήρως ε, εκδημοκρατισμένες χώρες, χάρη και στην ε, ανοιχτό χαρακτήρα που έδειξαν τότε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν υπάρξει θέμα, υπάρχει περιθώριο αναστολή τη συμφωνία. Ελπίζουμε όμω ποτέ να μην χρειαστεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Από του πράσινου το λόγο έχει η κυρία Στρίκ. Εν συντομία, Πρόεδρε, εξέφρασα κάποιε ανησυχίε ε, γενικά. Κοιτώντα τη συμφωνία επανεισδοχή με τη Λευκορωσία, για την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπιτανόφ. Εξαιρετική συνεργασία. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Η συμφωνία δεν ε, ε, υποχρεώνει τα κράτη να επιστρέψουν καταρχά του ανθρώπου στη χώρα προέλευση. Εδώ πέρα δεν υπάρχει οποιαδήποτε δίκλυντα ασφαλεία, ούτε υπάρχει υποχρέωση να χρησιμοποιούνται αυτέ οι επίσημε συμφωνίε. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιείται η ανεπίσημη συμφωνία, η ανεπίσημη διαδικασία. Και επίση υπάρχει και η επιταχυμένη διαδικασία, η οποία όμω είναι λίγο πιο επικίνδυνη σε ό,τι αφορά τι δικλείδε ασφαλείας. Να πούμε από πλευρά ε, του Κοινοβουλίου. Το πεδίο τη εντολή πλέον ορίζεται από το Συμβούλιο και μόνο. Αυτό το ορίζει η συνθήκη, αλλά θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αφήσει το Κοινοβούλιο να συμμετέχει από τη φάση της εντολής. Είπατε ότι ήδη υπάρχει διαδικασία χορήγηση ασύλου. Να πω όμω ότι οι συμφωνίε επανεισδοχή και οι ανεπίσημε αυτέ συνεργασίε έχουν ως στόχο να αποτρέπουν την ε, παράνομη μετανάστευση για να ενισχύονται οι έλεγχοι στα σύνορα και να μπορέσουν ε, οι άνθρωποι να περάσουν μέσω τη χώρα διέλευση ε, εκεί που χρειάζεται. Και εδώ λοιπόν επισημαίνουμε τι συνέπειε που θα είχε για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τέτοια άσκηση. Ο κύριος Φοντρόσο, δεν τον βλέπω εδώ από πλευράς του ID θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Για να ακούσουμε την κυρία Βυσνιεύσκα από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ECR υποστηρίζει τη Συμφωνία Επανεισδοχής καθώς και τη Συμφωνία Διευκολύνσεων για τις θεωρήσεις. Για μας είναι θετικό το πολιτικό μήνυμα το οποίο προσταλείται στη Λευκορωσία. Θέλουμε να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε τις ε, σχέσεις μας με τη χώρα αυτή, να καταστήσουμε και την ανθρώπινη επαφή πιο εύκολη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βιτάνοφ και τον κύριο Χου για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος από την ΚΟΕ η κυρία Ρέγκο. Δεν την βλέπω όμως στην αίθουσα. Θέλει να πάρει κανείς το λόγο εξ ονόματος της Γκουε. Όχι. Ο κύριος Μπράιερ είναι ο εισηγητής για το δεύτερο θέμα, το θέμα των διευκολύνσεων. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Yes, uh, thank you very much. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το, η Λευκορωσία είναι μια δικτατορία. Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη εκεί η που συνεχίζει να εφαρμόζει τη θανατική ποινή, η οποία εκτελείται μάλιστα με πυροβολισμό στο κεφάλι. Γνωρίζω, το γνωρίζετε. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένει κακή, χωρίς βελτιώσεις να παρατηρούνται. Αυτό συνεχίζει να αποτελεί ε, ανησυχία. Υπάρχουν, έχουν, ε, ε, εφαρμοστεί ακόμα, έχουν εφαρμοστεί ακόμα περισσότερες περισσότεροι περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να σιωπήσουν οι αντιφρονούντες. Έχουμε το Human Rights Watch το οποίο έχει καταγγείλει αυτές τις παραβιάσεις, έχει, κατα... έχει καταγγείλει αυθαίρετη κράτηση δημοσιογράφων, ε, καθώς επίσης και κράτηση ανθρώπων που διαμαρτύρονταν για το περιβάλλον. Ειρηνικά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ και ελπίζω ότι η Συμφωνία Απελευθέρωσης του Καθεστώτος Θεωρήσεων θα βοηθήσει να ανοίξει και να μετασχηματιστεί η χώρα αυτή και θα βοηθήσει και τη δουλειά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα αντιταχθούμε σε αυτή τη συμφωνία απελευθέρωση των θεωρήσεων, αλλά πρέπει να απαιτήσουμε ξεκάθαρα από τη Λευκορωσία να ε, σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αρχές της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε. Νομίζω ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις των σκιωδών. Κυρία Παριάτ, μιλάμε για το καθεστώς της Λευκορωσίας. Είναι διαβόητο το καθεστώς αυτό. Δεν υπάρχει σεβασμός για τη δημοκρατία, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρόεδρος είναι στη θέση του από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και δεν τον κουνάει κανείς. Επομένως, είναι ανησυχητική κατάσταση. Καταλαβαίνουμε και συμφωνούμε ότι είναι σημαντικές οι συμφωνίες επανεισδοχής και θεωρήσεων, αλλά μιλάμε για το είναι Λευκορωσία. Κύριε Χουκ, κύριε Βίτανοφ, είστε σκιώδεις εισηγητές για αυτά τα δύο σχετικά ε, θέματα νομίζω θα ήταν λογικό να σας δώσουμε το λόγο, ξεκινώντας από εσάς κύριε Βίτανοφ. Ναι, πράγματι ως σκιώδης εισηγητής για το δεύτερο φάκελο, για το δεύτερο θέμα παίρνω το λόγο. Να σας θυμίσω ότι το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει την πολιτική αυτές οι δύο συμφωνίες πανεσδοχής και θεωρήσεων να πηγαίνουν μαζί. Αναφέρθηκαν ήδη τα στατιστικά είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό κατακεφαλήν ε, θεωρήσεων που δίνονται στο χώρο Σέγγεν και με τις μικρότερο αριθμό επανεισδοχών. Ε, αυξήθηκε ε, από 60 σε 80 ευρώ το τέλος πρόσφατα εξαιτίας του νέου κώδικα θεωρήσεων. Όμως τώρα με τη νέα συμφωνία θα μειωθεί αυτό το τέλος στα 32 ευρώ. Γι' αυτό το λόγο με τους συναδέλφους συμφωνήσαμε να προωθήσουμε αυτούς τους φακέλους στο δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί όσο περισσότερο καθυστερεί έγκριση από το Κοινοβούλιο, τόσο περισσότερο καιρό αναγκάζονται οι άνθρωποι να πληρώνουν αυτά τα υψηλότερα τέλη. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω την αξιολόγηση που κάνει ο κ. Χουκ. Συμφωνώ μαζί του ότι το να υπάρχουν διαπροσωπικές επαφές ε, βοηθάει στην ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων, επιστημονικών σχέσεων και άλλων. Κύριε Χουκ, σύντομα κι εγώ. Συμφωνώ με τον συνάδελφο. Είναι σημαντικό αυτά τα δύο θέματα να τα δούμε μαζί, γιατί είναι οι δύο δίωδοι. Οι θεωρήσεις είναι ένας νόμιμος τρόπος να επισκεφτεί κανείς τη Λευκορωσία ή να επισκεφτεί κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστρόφως η επανεισδοχή είναι αυτό που συμβαίνει αν υπάρξει πρόβλημα. Ε, Επομένω, είναι λογικό αυτά τα δύο να πηγαίνουν χέρι-χέρι και αντιστροφως η επανεισδοχη ειναι αυτο που συμβαινει αν υπαρξει προβλημα επομενως ειναι λογικο αυτα τα δυο να πηγαινουν χερι χερι και είναι ένας τρόπος να προστατεύονται και οι Ευρωπαίοι που επισκέπτονται σε ορισμένες περιπτώσεις στη Λευκορωσία. Είναι σημαντικό να έχουν ε, προστασία σε αυτές τις ε, επισκέψεις στον τρόπο με τον οποίο θα τους αντιμετωπίζει το κράτος της Λευκορωσίας. Υπάρχει και αυτή η διάσταση και είναι εξίσου σημαντική. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο κυρία Παριάτη σε εσάς πάλι για την δευτερολογία σας για να ολοκληρώσετε. Έχουμε καθυστερήσει γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα σημαντικό για το ηλεκτρονικό αποδεικτικό υλικό να συζητήσουμε. Να ακούσουμε λοιπόν και εσάς μετά τις παρεμβάσεις των εισηγητών και των σκιωδών. Κυρία Παριάτ, δεν θα μακρηγορήσω κι εγώ. Βεβαίως είναι εύλογες οι ανησυχίες που έχετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να το αναγνωρίσω. Βεβαίως η εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχών είναι με την αίρεση βεβαίως των υποχρεώσεων που έχει η Λευκορωσία υπό το διεθνές δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με την αρχή της μη επαναπρόθεσης. Από την άλλη, η Συμφωνία Θεωρήσεων έχει μια συγκεκριμένη αναφορά στο προήμιό της, το γεγονό ότι και τα δύο μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία του σεβασμού τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να επισημάνω ότι κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια αναφορά δεν έχουμε σε καμία άλλη συμφωνία θεωρήσεων που να έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουμε λοιπόν ότι μπορούμε να προωθήσουμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Αυτό μόνο ήθελα να προσθέσω στο πρωτολογία μου. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα που ακούσαμε και τα δικά σας σχόλια μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα, με μια μικρή καθυστέρηση. γιατί θα έχουμε την συζήτηση για το ηλεκτρονικό υποδεικτικό υλικό και άλλες συζητήσεις. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και καλή ε, επιτυχία στη νέα σας ιδιότητα. Είναι σίγουρο ότι θα συναντώμαστε και θα συνεργαζόμαστε πολύ συχνά. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Όπως είπα, έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε ένα ευαίσθητο θέμα που μας έχει μείνει από την προηγούμενη θητεία και πρέπει να επιταχύνουμε για να προλάβουμε. Παρακαλώ, ησυχία. Είναι πολύ σοβαρό, ε, νομοθετικό, πολύ σοβαρό το νομοθετικό ντοσχέ αυτό για την δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει. Την ε, τήρηση διαταγών και εντολών για την ε, τήρηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων με εισηγήτρια την κυρία Σίπελ. Έχουμε εδώ την πρόταση οδηγίας για εναρμονισμένους κανόνες για τους νομικούς συνηγόρους και για την τήρηση των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων ή evidence και οδηγία για νομικούς αντιπροσώπους. για να μπορούν να φέρουν τις αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικέ υποθέσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων. Κυρία Σίπελ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους Κιώδης για την στενή συνεργασία στο θέμα και στους άλλους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν με την υποβολή τροπολογιών. Για να θυμίσω τι έχει γίνει. Τέλη Νοεμβρίου λάβαμε 841 τροπολογίες για το προτινόμενο κανονισμό και άλλες 26 για την προτινόμενη οδηγία. Τον Ιανουάριο είχαμε και όλες τις μεταφράσεις. Εάν δούμε πόσες τροπολογίες υποβλήθηκαν από πόσους συναδέλφους και το όλο περιεχόμενο, δύο πράγματα είναι τελείω σαφή. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φάκελο αυτό, για το θέμα αυτό, ασχέτω πολιτική ομάδα και χώρα προέλευση. Αλλά γενικότερα υπάρχει μια ευρία πλειοψηφία που είναι υπέρ του να βρεθεί μια καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ των όσων ε, θέλουν οι διοικητικέ αρχέ και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για να το πω διαφορετικά, η ευρία πλειοψηφία ομάδων και συναδέλφων δεν υποστηρίζει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω έχει σκοπό έχει αυτή να δημιουργήσει ένα μηχανισμό που θα επιτρέπει στις αρχές ενός κατους μέλους να ζητήσουν απευθείας την αποκάλυψη και τήρηση όλων των ειδών στοιχείων από τους παρόχους των στοιχείων αυτών σε άλλο κράτος μέλος χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς καμία πληροφορία ε, προς τη χώρα που βρίσκεται ο πάροχος των πληροφοριών ούτε στη χώρα του θυγόμενου, του ενδιαφερόμενου προσώπου οπότε δεν υπάρχει και δικαίωμα ένστασης μομφής κατά της ε, ε, κατά του της αποκάλυψης. Ζητούμε λοιπόν την ε, δυνατότητα συμμετοχή του κράτου, όπου βρίσκεται αυτό που παρέχει τι πληροφορίε, τα αποδεκτικά στοιχεία, ή εκεί που αντιπροσωπεύεται, και κάποια, κάποιοι συνάδελφοι ζητούν την συμμετοχή του κράτου, όπου ο θυγόμενο, ο ενδιαφερόμενο ή ο δικαζόμενο έχει το, την έδρα του, ε, αυτό που είναι γνωστό τώρα σε αγγίλε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αυτό θα ε, χρειάζεται για ένα πολύ περιορισμένο αριθμό υποθέσεων. Εν γέννη, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στο άρθρο 82.1, το οποίο έχει να κάνει με την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Συμφωνούμε όλοι ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι ως λίθος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας όμως δεν μπορεί να εφαρμόζεται από πάνω προς τα κάτω, να επιβάλλεται δηλαδή και δεν μπορεί να είναι τυφλή αυτή η εμπιστοσύνη. Δεν ομιλώ μόνο για τους προφανείς, τους συνήθεις υπόπτους που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη, αλλά μιλάω για όλα τα κράτη-μέλη συνολικά. Και έχω μάλιστα πληροφορίες ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν κάπως ανησυχήσει με την εμπιστοσύνη που μπορεί να δείχνουμε προς όλα τα κράτη-μέλη ανεξαιρέτως. Επιπλέον, στο άρθρο 82.1 μιλάμε για δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει. Όμως, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει μια εντελώς νέα ερμηνεία από την αρχή ενό κράτου μέλου προ μια ιδιωτική εταιρεία ή φορέα προ ένα άλλο κράτο μέλο. Εδώ λοιπόν πρέπει να έχουμε υπόψη ότι παρά τις εντατικέ μας προσπάθειες πέρσι για να εναρμονίσουμε τα συστήματά μας, η ποινική δικαιοσύνη και τα συστήματά της είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους από χώρα σε χώρα. Διαφορετική, ε, ε, διαφορετικός ορισμός εγκλημάτων, διαφορετική επιβολή ε, ποινών και κυρώσεων, διαφορετικές δυνατότητες για τις διοκτικέ αρχές, διαφορετικά συστήματα για την συλλογή και τήρηση αποδεκτικών στοιχείων. Γι' αυτό η, παραδοσιακή ευθύνη που αναλαμβάνουν οι κρατικέ αρχές δεν μπορεί να πηγαίνει προς τις ιδιωτικέ εταιρείε. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε ένα μηχανισμό κοινοποίηση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορούν να αρνηθούν, να αναγνωρίσουν ή να εκτελέσουν τέτοιε εντολέ για, για πολίτε που βρίσκονται στην επικράτειά του βάσει συγκεκριμένων ε, αιτίων. Οι ιδιοκτικέ αρχέ θα πρέπει να γνωρίζουν και τι νέε τάσει των ε, εγκληματικών ε, ενεργειών, είτε στην επικράτειά του είτε σε άλλε χώρε. Βλέπω ότι είναι πολλοί συνάδελφοι που συμμερίζονται την άποψη αυτή και χαίρομαι γι' αυτό. Ταυτόχρονα όμω ισχύει ε, ότι για να σχεδιαστεί σωστά ένα τέτοιο μηχανισμό και να βρούμε τη σωστή, το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ των όσων επιθυμούν οι διοικητικέ αρχέ και τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εκεί ακριβώ το σημείο αυτό αποκλίνουν οι απόψει μα. Ο μηχανισμό κοινοποίηση και η διαδικασία εφαρμογή του πάνε χέρι-χέρι με άλλε τροπολογίε που προτείναμε κάποιοι από εμά ό,τι αφορά την τήρηση ε, αποδεκτικών στοιχείων, τι ε, τη διάρκεια τήρησης, ε, την ε, εκδίκαση της υπόθεσης και ούτω καθεξής. Επίσης, η κοινοποίηση και ενημέρωση μιας αρχής και ασφαλής δίωδη για τη μεταφορά των στοιχείων είναι θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους. Όλα αυτά βρίσκονται επιτάπητος, έχουν όλοι διαφορετικές απόψεις. Θα σταματήσω εδώ προς στιγμή και αφήνω το λόγο στους και εισηγητές για να πούνε εκείνοι τις δικές τους απόψεις και τις τροπολογίες τους, να παρουσιάσουν τις τροπολογίες τους. Ευχαριστούμε κυρία Σίπελ για την παρουσίαση αυτού του ευαίσθητου θέματος. Είναι δύσκολο το ντοσιέ. Ανακεφαλαίωσατε τις ε, διαφορές μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου αρκετά καλά. Γι' αυτό και προέκυψαν τόσο πολλές τροπολογίες και γι' αυτό ε, καλό θα ήταν να ακούσουμε τους κοιόδης συζητητές για να δούμε αν υπάρχει κάποιο περιθώριο ώστε να υπερπηδήσουμε τις δυσκολίες που είχαμε τώρα. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον σκιώδη του ΕΛΚ, τον κύριο Λένερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σκιώδης μας είναι ο κύριος Μέλου, αλλά δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Οπότε μου ζήτησε να σας παρουσιάσω μερικές από τις ιδέες του. Έχει υποβάλει 94 τροπολογίες. Και όπως είπε και η συγγήτρια, Σκοπό ήταν να βρεθεί το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ του να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό, αλλά να προστατεύουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα ταυτόχρονα και να υπάρχει και νομική βεβαιότητα για όσου παρέχουν ε, τι σχετικέ πληροφορίε. Ένα σημαντικό σημείο για τον κύριο Μέλλο μέσα από τι τροπολογίε του είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί η διάρκεια τήρηση των στοιχείων από τρία σε δύο χρόνια στο γαλλικό δίκαιο, α πούμε, έχουμε τιμωρία για την παιδική πορνογραφία δύο χρόνια και εδώ η τήρηση ηλεκτρονικών στοιχείων είναι σημαντική για τέτοια σοβαρά ε, ε, εγκλήματα. Τρία χρόνια, λοιπόν, είναι το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ της ε, αναλογικότητα και των επιθυμιών των διεκτικών αρχών. Ο εισηγητή θέλει λοιπόν συνολικά θα επιθυμούσε το όριο των 5 ετών, αλλά για σοβαρά έγκληματα, όπω να είναι κάποιο ε, μέλο συμμορία ε, στο Βέλγιο ή την υποστήριξη δημοκρατικών οργανώσεων στη Γερμανία. Επίση, τα ευρωπαϊκά εντάλματα έρευνα και η τήρηση σχετικών ε, στοιχείων για τέτοια εγκλήματα με τον κίνδυνο ατιμορρησία για σοβαρά εγκλήματα είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη για το, για το σύστημα κοινοποίηση. Και μόνο για τι ευρωπαϊκέ δικαστικέ εντολέ, για τα στοιχεία συναλλαγών και εκεί όπου οι αρχές έκδοσης έχουν ε, λόγους να πιστεύουν ότι δεν κατοικεί στη χώρα έκδοσης ε, ο ενδιαφερόμενος, τότε θα πρέπει η αρχή επιβολής του νόμου να μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα με δυνατότητα ένστασης 10 μέρες και η τεκμηρίωση της ένστασης να είναι ε, ένα περιορισμένο σύνολο κριτηρίων. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα υποβολής περαιτέρω, για περαιτέρω πληροφορίες. Ο εισηγητή εδώ έχει μια ελαφρώς διαφορετική πρόταση, συστηματική συμμετοχή των αρχών του κράτους μέλους που θα πρέπει να εκτελέσει την εντολή. Θα πρέπει να λαμβάνεται ξεχωριστά απόφαση για κάθε εντολή ακόμα και για, αρχή, για ε, έτοιμα τήρησης ή αποστολής δεδομένων, ο κύριος, Νένο, ο κύριος Μέλου θεωρεί ότι η διαδικασία θα είναι πιο περίπλοκη από αυτή που τώρα υπάρχει. Οπότε, εφόσον δεν υπάρχουν νομικοί αντιπρόσωποι, ε, στην επικράτεια, όπω συμβαίνει λόγω χάρη στην Ιρλανδία, κατά, κάθε χρόνο θα υποβάλλονται εκατοντάδε αιτήματα και θα, αυτό θα βαρύνει ιδιαίτερα τι αρχέ. Επίση, μια σύντομη προθεσμία απάντησε 8 ώρε για τα σχετικά αιτήματα σε σχέση με τι 6 που προτείνει η Επιτροπή και τις 24 που προτείνει η συγγήτρια και για την τήρηση τη Ευρωπαϊκή εντολής. Ο κύριος Μέλο λέει ότι ε, περιμένει να δει τι συμβαστικέ τροπολογίε του Δενού συντομότερα και, για να τονίσει, και τονίζεται για το ΕΛΚ ότι θα πρέπει να χωρίσουμε τα στοιχεία σε τέτοιε κατηγορίε ώστε οι διοικητικέ αρχέ να μπορούν να τα εντοπίσουν αναλόγως για να ξέρουν αν θα ε, κάνουν αναλόγως και τις έρευνες για τους δράστες και αυτούργους και να δούμε αν ικανοποιούνται προτεραιότητες που έχει θέσει το ΕΛΚ. Πρέπει όντως να επιταχύνουμε για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό έγκλημα και να έχουμε ταχές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των ε, σοβαρών εγκλημάτων. Όπως είπατε λοιπόν Πρόεδρε, πρέπει να βρούμε κάποιο περιθώριο, αλλά θα πρέπει κάποιο να κινείται για να υπάρξει το περιθώριο αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Κονέ, ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω την εισηγητρία την κυρία Σίπελ για τη δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό και τους υπόλοιπους κοιόδης και τους συναδέλφου που έκαναν πραγματικά τόσες, ε, κατέθεσαν τόσες πολλές τροπολογίες. Είναι μεγάλο ο όγκο τη δουλειά. Θεωρώ ότι αυτό το εργαλείο γενικά είναι υπέρ τη Ευρώπη. Και αφορά βασικά θέματα εμπιστοσύνη. Πόσο εμπιστευόμαστε τις αρχέ άλλων κρατών μελών να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Και η πρόταση αυτή επίση έχει να κάνει και με την ενιαία αγορά. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τι συνέπειε μια πραγματικά ενιαία αγοράς. Σε ό,τι αφορά ένα επιπλέον εργαλείο Συμφωνώ για το επιπρόσθετο εργαλείο που χρειάζεται σε σχέση με το ΙΑΟ. Και επίση συμφωνώ σε ό,τι αφορά τι ανοιχτέ αγορέ για τι ψηφιακέ υπηρεσίε. Συμφωνώ εκ παραλλήλου και με του σοσιαλδημοκράτε και με την εισηγήτρια ότι σε κάποιε περιπτώσει το εργαλείο αυτό ενδεχομένω να τέχει κατάχρηση για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρειάζεται κάποια δικλίδα ασφαλεία. Συμφωνώ και με του πράσινου και με την ΚΟΕ ότι το σύστημα κοινοποίηση από μόνο του δεν θα αποτελέσει την ε, σωστή δικλίδα ασφαλεία. Και προτείνω λοιπόν τροπολογίε οι οποίε θα ενσαματώσουν ε, και δικλίδε ασφαλεία και θα επιτρέψουν να λειτουργήσει αποτελεσματικά το εργαλείο αυτό. Θέλω να υπάρξει συμβιβασμό μεταξύ των μεγάλων ε, ομάδων που είναι υπέρ τη Ευρώπη. Είτε σκοπός είναι να εντοπιστεί ένα άτομο, είτε επίσης Μα απασχολεί κάτι παραπάνω πέρα από την τοποθεσία του σερβερ ή κατά πόσον πρόκειται για χώρα, ε, είτε πρόκειται για τα χώρα που υπόκειται στη διαδικασία του άρθρου 7. Ε, πιστεύω ότι αυτές οι μεταφορές θα επιτρέψουν τη γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων σε ό,τι αφορά και το, την εξαίρεση της ε, του δικαιώματο αίτηση ε, πληροφοριών ε, για προστατευμένα επαγγέλματα, όπω του δημοσιογράφου. Θεωρώ ότι αυτό θα αποτελέσει σωστά, σωστή ισορροπία. Επίση, είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι θα πρέπει να υπάρξει μια υποδομή IT η οποία θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των παρόχων και των αρχών, όπως είπε και η συγκήτρια. Πιστεύω ότι χρειάζεται εδώ να υπάρχουν ασφαλείς δίωδοι και απαραίτητη πιστοποίηση τον ε, επαλήθευση των ε, ετοιμάτων. Θεωρώ ότι με αυτά μπορούμε να πετύχουμε μια ευρεία συμφωνία στο Κοινοβούλιο και να προσεγγίσουμε το Συμβούλιο, να έχουμε υπόψη μας ότι θα είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις και τρεμερείς διάλογοι και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί και να υπάρχει σωστή πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Προσβλέπω λοιπόν ε, στη συνεργασία και στην εξέβρεση συμφωνιών και συμβιβασμών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαγκορίνης και από τους Πράσινους. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον ε, συνεισηγητρία για την ε, ακούραστη δουλειά που έκανε. Μεγάλο θέμα. Και προφανώς έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ε, η κυρία Σίπελ. Υποστηρίζουμε γενικά τις γενικές γραμμές της πρότασης. Υποστηρίζουμε και όλος ιδιαίτερος τη συμπερίληψη των διατάξεων για τους νομιμούς εκπροσώπους στον κανονισμό. Από αυτόν συμφωνούμε. Και τη γενική κατεύθυνση υποστηρίζουμε. Αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφάνεια μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα για τους εμπλεκόμενους φορείς, για τις αρχές, σε ό,τι αφορά διάφορα διαδικαστικά και διάφορες ε, διαδικασίες. Κατάσχασα, έχουμε τις ε, κατηγορίες δεδομένων, όπως προτείνονται από την κυρία εισηγήτρια, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των ε, συνδρομητών κτλ. Αλλά οι ορισμοί περιεχομένου από την σχετική νομοθεσία έχει περιοριστεί σε σχέση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Θα θέλαμε λοιπόν να διευκρινίσουμε αυτό το σκέλος. Ένα άλλο θέμα είναι ο ορισμός του εκτελόντος κράτους. Ε, προτείνουμε να μπει μια σταδιακή ρήτρα για την ευκρίνηση των ε, ορισμών εκεί που ορίζονται καταρχάς ε, τα δεδομένα. Μετά να κοιτάξουμε τη βασική, ε, το βασικό ε, την έδρα τη εταιρεία. Και εκεί, αν εκεί τα πράγματα είναι εντάξει, να κοιτάξουμε και τις άλλες εγκαταστάσεις της εταιρεία σε άλλα κράτη-μέλη ενδεχομένω. Και μόνο ως τελευταία ίστατη λύση να κοιτάξουμε το θέμα ε, του νομιμού αντιπροσώπου. Αυτό περιλαμβάνεται και στον επιστολή που υπευλήθηκε στη ΣΥΠΑ σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία, όπου παρουσιάστηκε πραγματικά ακριβώς αυτή η πρόταση από πλευρά μας. Θέλουμε να διευκρινίσει επίσης ε, τι αρμοδιότητες ε, κοινοποίησης έχουν οι αρχές στον διασυνοριακό μηχανισμό. Προτείνει η συγγήτρια η εκτελεστική αρχή να έχει τη δυνατότητα παρέμβαση σε κάποιο χρονικό διάστημα συγκεκριμένο. Εμεί ξέρουμε πώ λειτουργούν οι αρχέ και ξέρουμε πόσο κατακλυσμένε είναι. Ευχαριστώ τον συνάδελφο από το ΕΛΚ που το ανέφερε. Ξέρουμε πόσο φόρτο εργασία έχουν οι δικαστικέ αρχέ. Όπω και να έχει λοιπόν, δεν θα έχουν τη διάθεση ούτε το χρόνο να κάνουν την κοινοποίηση εντό του πλαισίου αυτού. Θα πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουμε σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρεια. Και σε ό,τι αφορά τον προορισμό σε χώρε άρθρου 7, θα εξαιρούσε τι άλλε χώρε. Αυτό το όριο είναι υπερβολικά υψηλό, γιατί έχουμε προβλήματα δικαστική εμπιστοσύνη. Το ακούσαμε και στο Ζάγκρεπ την προηγούμενη εβδομάδα με του υπουργού δικαιοσύνη. Η δικαστική εμπιστοσύνη δεν περιορίζεται σε δύο χώρε εκεί που υπάρχει η διαδικασία του άρθρου 7 θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο ευρέω για το πώ θα εξασφαλίσουμε και θα κατοχυρώσουμε σωστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χρειάζεται λοιπόν ε, ρετή απόφαση της ε, εκτελεστικής εξουσίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά την προστασία προς τους δημοσιογράφους μέσω του ελέγχου αυτού. Προτείνουμε να αποφύγουμε τη διαγραφή υλικού, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και οι, οι εταιρείε δεν θα πρέπει να είναι η πρώτη γραμμή προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Συμφωνούμε από, αυτό, Αν θεωρηθεί ότι ε, ένα αίτημα είναι καταχρηστικό, κατά εξοχήν, θα πρέπει να είτε να ζητήσουν πιο πολλέ πληροφορίε πρωτού ληφθεί η απόφαση ή να στραφούμε προς την εκτελεστική εξουσία. Για τους λόγους τώρα μη αναγνώριση και μη εκτέλεση αποφάσεων και τιμάτων, ε, μη εκτέλεση εντάλματο. Εδώ χρειάζεται πιο πολλά στοιχεία από το ευρωπαϊκό ένταλμα και να επιτρέπεται από μια αρχή να ζητά δεδομένα. Εδώ αυτό είναι βασικό στοιχείο. Θεωρούμε σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό αποδεικτικό υλικό, πρόκειται για μία εξαίρεση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Ε, ζητάμε λοιπόν εξέταση του ευρωπαϊκού εντάλματος, προκειμένου τελικά να ενταχθούν στο πλαίσιο του EIO και τα, το αποδεκτικό υλικό αυτό. Μία τελευταία τώρα σημείωση όχι τόσο κρίσιμη σημασία, αλλά παρόλα αυτά καλό είναι να αναφερθεί. Μιλάμε για κρίσιμε υποδομές ε, και αυτό αποτελεί κριτήριο παραδεκτότητας. Εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό και αυτό το έχουμε συζητήσει με του δικαστέ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τι γίνεται αν η παραδεκτότητα αποδεκτικού υλικού στην χώρα εκτέλεσης και στη χώρα που ζητά τα δεδομένα είναι διαφορετικέ οι όροι αυτοί. Αν δηλαδή τα στοιχεία αυτά, ε, τα απαιτητικά στοιχεία αυτά είναι παραδεκτά στη μία χώρα και όχι στην άλλη. Εδώ θα πρέπει να ε, αφιερώσουμε μία τροπολογία για να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο αυτό. Άρα, έχουμε τι διαδικασίε του άρθρου 7, έχουμε την έλλειψη δικαστική εμπιστοσύνη μεταξύ διαφορών χώρων και στο παρόν σημείο δίνουμε μία πρόταση που θα δώσει στις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης εμπιστοσύνης ε, πολύ ευρεία δικαιώματα και αρμοδιότητες. Αυτό πραγματικά ας μην το κάνουμε, ας το σκεφτούμε καλά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δεδομένα αυτά βρίσκονται σε κάποια χώρα, ενώ ε, ο δράστης είναι σε άλλη χώρα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα στοιχεία. Ας δούμε τι γίνεται, για παράδειγμα, στη Σλοβακία. Μιλάμε για το μοναδικό, ε, τη μοναδική εταιρεία ανεξάρτητων ε, δεδομένων. Και πού αποθηκεύονται όλα αυτά τα στοιχεία, μα όχι στη Σλοβακία, εκτός Σλοβακίας. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι τυχαίο. Ας σκεφτούμε λοιπόν αυτά πριν αποφασίσουμε για το φάκελο αυτό. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του ID. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους σκιώδες για τη δουλειά που κάνουμε για το θέμα αυτό που είναι ιδιαίτερα τεχνικό και περίπλοκο, αλλά έχει μεγάλη σημασία γιατί θα έχει μεγάλες πρακτικές συνέπειες για την δίωξη εγκλημάτων και την αναχέτηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το κείμενο της εισηγήτριας αλλάζει σοβαρά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμένα, εμάς μας φαίνεται καλύτερα εξισορροπημένη. Διαφέρει σε πολλά σημεία, όπως τις διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων. Γι' αυτό έχω υποβάλει 16 τροπολογίες, οι οποίες σκοπό έχουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα όσων προβλέπονται, αλλαγή των όρων για την τήρηση των δεδομένων, αλλά και διατάξεις που θα επιτρέπουν να λάβουμε περισσότερο υπόψη την ποικιλομορφία των δικαστικών συστημάτων. Κάποια σημαντικά σημεία για μας τα ανέφερε και ο συνάδελφος του ΕΛΚ, γι' αυτό δεν θα τα επαναλάβω. Όμως θέλω να επισημάνω ότι η διαδρομή της κοινοποίηση γίνεται πολύ πιο αυστηρή από την αρχική πρόταση και περνά τα, ξεπερνά τα όρια του λογικού, διότι οι αρχές θα πρέπει να μπορούν ε, ταχαίως να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία που χρειάζονται. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε για να βρούμε συμβαστικέ λύσεις ώστε να διευκολύνουμε την εργασία των δικαστικών ε, αρχών σεβόμενοι πλήρω τα, δικαιώματα, τα δικαιώματα των πολιτών. Για τις ηλεκτρονικές εξελίξεις και την προστασία των θεμελιδών δικαιωμάτων επίση. Υπάρχουν πολλά σημεία του ντοσχέ που θα πρέπει να δούμε την, το συγκερασμό των δύο θεμάτων. Και για τα όρια των ποινών, όπως είχα πει και σε προηγούμενες συζητήσεις, θεωρώ ότι είναι καλύτερη η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, ελάχιστος χρόνος ε, τήρησης τριών χρόνων ε, από τα πέντε χρόνια, καλύτερα από τα πέντε χρόνια που προτείνει η συγγήτρια. Θεωρώ μάλιστα ότι πολλές χώρες θα βρίσκονταν εκτός του πεδίου εφαρμογή αυτού του εργαλείου για ορισμένα αδικήματα ή εγκλήματα όπου οι ηλεκτρονικές αποδείξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο. Το stalking δηλαδή, η παρενόχληση που συστηματική παρενόχληση στην Ιταλία τιμωρείται με τέσσερα χρόνια, Όμω εκεί δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά στοιχεία. Εδώ λοιπόν χρειάζεται ένα εργαλείο το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει γρήγορα, αλλά να είναι και δραστικό και αποτελεσματικό. Θα πρέπει οι διαδικασίε να σέβονται τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων, ακόμη και όσων συμμετέχουν απλώ στη διαδικασία, τη. Ε, στα αποδεικτικά στοιχεία. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε με προσοχή τις τροπολογίες όπου ε, τελικά καταλήγουμε σε μια υπέρμετη προστασία των ατομικών δικαιωμάτων αλλά περιορίζοντας την δραστικότητα και των ε, εντολών τήρησης, συλλογών, τήρησης στοιχείων και το πόσο καιρό πρέπει να διατηρούνται. Δεν βλέπω εκπρόσωπο του ECR. Η κυρία Έγκστρα του Ινγκουε. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να συλλέγουμε και να μεταφέρουμε τόσο πιο, όσο πιο γρήγορα γίνεται τα στοιχεία αυτά, αλλά να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι το θέμα αυτό που ανέφερε ένας συνάδελφος από το Renew, να υπάρχει και εμπιστοσύνη. Είναι θέμα εμπιστοσύνη το θέμα αυτό. Πόσο σίγουροι είμαστε σε ό,τι αφορά μεταφορά στοιχείων σε άλλα κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα θεμελιώδη δικαιώματα κάποιων ατόμων και τα προσωπικά τους δεδομένα. Και δεν μιλάμε μόνο για τις χώρες του άρθρου 7. Ε, φυσικά όλος ο είναι το θέμα αυτό σχετικό για τις χώρες αυτές του άρθρου 7. Και ξέρουμε πόσο ε, μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα και επίμονα τα προβλήματα αυτά και πόσο ανίσχυροι είμαστε ουσιαστικά. Είμαι πραγματικά διστακτική σε ό,τι αφορά ε, το σύνολο του εργαλείου αυτού, του μέσου αυτού. Αν θέλουμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε και καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα τίθεται θέμα συμβασμού, θα πρέπει να ε, εξετάσουμε δελεχώς το θέμα των θεμελιδών δικαιωμάτων. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι από τους πράσινους, από του Renew και η συγκητρία να πω μόνο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα τριπλό σενάριο. Αν δείτε εμ, τις τροπολογίες μας, μιλάμε για, για εντολές διατηρήσεις οι οποίε ε, θα πρέπει να τηρηθούν. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί εδώ σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που υπάρχουν. Είναι περιορισμένε ε, για να μπορεί κανείς να αντισταθεί στο αίτημα χορήγησης στοιχείων, αλλά οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τους παραδοσιακούς λόγους άρνησης χορήγησης στοιχείων σε ό,τι αφορά ε, τις εντολές ε, παραγωγής και των ε, στοιχείων συνδρομητών και το data for traffic και content data. Όλα αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να διακριθούν καλύτερα το ένα από το άλλο, να γίνει καλύτερη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα δεδομένα συνδρομητών, subscriber data. Πιστεύουμε ότι και θα πρέπει να αποσταλθούν από τις αρχές και στους συνδρίες. Και όπως είπε η συγγήτρια, η, η αρχή εκτέλεση θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει απόφαση. Αν δεν ληφθεί η απόφαση όμως εντός συγκεκριμένη προθεσμίας, οι πάροχοι θα πρέπει να μπορούν να αποστέλουν τα στοιχεία που ζητούνται διαφορά τώρα μεταξύ δεδομένων traffic και content. Αυτά θα πρέπει να μπορούν να αποστέλλονται στην ε, αρχή εκτέλεση. Σε αυτή την ειδική περίπτωση, λοιπόν, θέλουμε να έχουμε πιο ε, καλέ εγγυήσει από αυτέ που προβλέπονται στο σχέδιο κειμένου. Η executing authority, η αρχή εκτέλεση, θα πρέπει να λαμβάνει απόφαση. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την εντολή και να μπορεί να αρνείται σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει ενδεχόμενη ή ενδυνάμει παραβίαση δικαιωμάτων. Γιατί θεωρώ ότι η ενδυναμει παραβιαση δικαιωματων γιατι θεωρω οτι η διδικοποιηση τη εργασία αυτή περιέχει πολλού κινδύνου. Και να πω και κάτι άλλο για τι τρίτε χώρε σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση με το δίκαιο και την νομοθεσία τρίτων χώρων. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Προσπαθήσαμε να κάνουμε πιο αυστηρές ε, τις ε, υποχρεώσει για τι αρχέ των τρίτων χωρών, όπω ζήτησε και το EDPS. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει κάποια ρύθμιση περαιτέρω. Δεν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε καταστάσει ε, που θα εκθέσουμε τα στοιχεία μα σε αμερικανικέ ε, υπηρεσίε. Αυτό αποτελεί μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που δήλωσαν το ΕΛΚ και για άλλε ομάδε και θα πρέπει όλα αυτά να τα συζητήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Ναι. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πώς βλέπει τα πράγματα αυτά σε αυτό το θέμα και η Επιτροπή. Κυρία Σφέτε, έχετε το λόγο και μετά θα ξαναδώσω στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτιμούμε ιδιαίτερω τι προσπάθειε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πλευρά τη Επιτροπή να προσπαθήσει να προωθήσει το φάκελο αυτό και να τον εξετάσει σοβαρά. Και η όποια λύση θα βρεθεί στο τέλος θα πρέπει να είναι και αποτελεσματική και να προστατεύει αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέντε σημεία θα ήθελα να επισημάνω. Πρώτον, να υπενθυμίσω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις όταν έχουμε ηλεκτρονικό αποδεικτικό υλικό ε, που το ζητούν οι ιδιοκτικές ή δικαστικές αρχές, ο χρήστης ήθεστε να βρίσκεται στο, στη χώρα εκείνη που εκδίδει το αίτημα. Αυτό ισχύει στο 94% των περιπτώσεων. Επομένως, πρόκειται κατά κύριο λόγο για εθνικές ε, περιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από τις περιπτώσεις, κύριε, για παράδειγμα, που ζητείτε έρευνα κατοίκων, για τις οποίες έχουμε ήδη μηχανισμούς συνεργασίας, όπως την ε, Ευρωπαϊκή Εντολή Δικαστικής Συνεργασίας. Εδώ ε, έχουμε ένα, μια διαφορετική συζήτηση ένα εργαλείο που διαφέρει από τα παραδοσιακά ε, διοκτικά και ερευνητικά εργαλεία. Δεύτερον, αυτή η συζήτηση για την κοινοποίηση και για την αρχιτεκτονική του συστήματος που εισάγει ο κανονισμός για την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Θα ήθελα και πάλι να επιθυμίσω ότι η όποια λύση θα πρέπει να βελτιώσει την πρόσβαση στα ηλεκτρονικό αποδεικτικό υλικό, όχι να, το κάνει, να κάνει αυτή την πρόσβαση πιο επαχθή. Επομένως θα πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε λύσεις οι οποίες να είναι πιο περίπλοκες από, αυτές, από, την δυνατότητα, από τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Έρευνας. Υπ' αυτή την έννοια, διαπιστώνουμε ότι ναι, καμία από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τις προθεσμίες που έχει θέσει η πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή για την διάκριση μεταξύ επιγουσών υποθέσεων και άλλων, και το καλωσορίζουμε αυτό γιατί το όποιο σύστημα θα πρέπει να, είναι, ε, να μπορεί να λειτουργήσει και με αυτές τις προθεσμίες. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες οι οποίες προτείνουν να αυξηθεί το όριο για, το περιεχόμενο, για τα ε, στοιχεία θέσης των συναλλαγών, transaction, ή να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην περιορίσουμε υπερβολικά το πεδίο εφαρμογής αν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα νομοθέτημα το οποίο να έχει προστιθέμενη αξία. Οποιοδήποτε, οποιοδήποτε περιορισμός του πεδίου εφαρμογή σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιες περιπτώσεις υποθέσεων, κάποιες ε, διοκτικέ ε, ενέργειες τις οποίες θα δυσκολέψουμε. Θα πρέπει να μην το ξεχάσουμε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τι κατηγορίες δεδομένων, από την πλευρά εκείνων που ασχολούνται στην πράξη με τα θέματα αυτά μας ζητούν να έχουν ευκολότερη δυνατό, να διευκολύνουμε μάλλον τη δυνατότητά τους να ταυτοποιούν τα πρόσωπα, γιατί αυτό είναι το πρώτο στάδιο σε οποιαδήποτε ιδιοκτική ε, διαδικασία. Αυτό ε, έχει σχέση και με τα δεδομένα συνδρομητή, αλλά και με τα δεδομένα πρόσβασης, subscriber και access. Τέλος, δεν είναι τόσο πολιτικό το θέμα, αυτό που θα σας επισημάνω, αλλά περισσότερο νομικού χαρακτήρα. Έχουμε προτείνει ε, δύο ε, νομοθετήματα και κανονισμό και οδηγία για νομικούς λόγους. Αυτό είναι, αυτό είναι σημαντικό. Επομένως, δεν θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να μην έχουμε οδηγία και να ενσωματώσουμε όλα όσα τώρα είναι στην οδηγία σε κανονισμό. Αυτό θα δημιουργήσει νομικά προβλήματα, δεν είναι εφικτό. Τώρα, όσον αφορά το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγή δεδομένων, είναι αυτό, κάτι το είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίζει το ευρωπαϊκό ένταλμα ερευνά. Θα μπορούσαμε να σα παρουσιάσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμή για το σύστημα αυτό στο Κοινοβούλιο, αν σα ενδιαφέρει, γιατί θεωρούμε ότι ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα. Έχει υπάρξει δηλαδή μια δουλειά στη δημιουργία ενό ασφαλού συστήματο ανταλλαγή δεδομένων. Προσβλέπουμε στην αποτελεσματική συνεργασία με το συνομοθέτη ώστε να βρεθεί συμβιβαστική λύση σε αυτό το σημαντικό φάκελο και έχουμε και εμεί ένα ερώτημα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, τι προβλέπετε για τα επόμενα βήματα. Ευχαριστώ, θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα με βοηθούσε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αυτή την παρουσίαση που μας πρότεινε για τα ασφαλή κανάλια ανταλλαγής δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, να δούμε πώς αυτή η νομοθεσία θα εφαρμοστεί στην πράξη. Θα έρθω τώρα σε όλα αυτά τα επιχειρήματα που παρουσίασαν οι σκιώδεις εισηγητές. Βλέποντας και τις τρομπολογίες ε, και την επιχειρηματολογία, είναι ξεκάθαρο ότι το θέμα είναι σημαντικό και από τεχνική και από νομική άποψη και επίσης σχετίζεται με πολύ ευαίσθητα θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έχουν αντιμετωπίσει το ζήτημα με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ένα από τα κυριότερα θέματα στη συζήτηση αυτή που ακούσαμε είναι ότι υπάρχουν ορισμένε πολιτικέ ομάδε οι οποίε θέλουν να δημιουργηθεί μια πολύ ισχυρή διαδικασία κοινοποιήσεων, η οποία μάλιστα να δημιουργεί και ε, ε, ε, την δυνατότητα παύση τη ανταλλαγή των δεδομένων για όλε τι κατηγορίε. Εγώ προ... και προτείνεται εντός του χρονικού ορίου που προτείνει η Επιτροπή, εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, να υπάρχει κοινοποίηση. Σε ορισμένη περιπτώ... μάλιστα έχουμε και δύο πολιτικέ ομάδε οι οποίε ζητούν ε, να, να... να χρειάζεται να γίνει θετική έγκριση ε, πριν να παρουσιαστούν αυτά τα δεδομένα. Εμείς ζητούμε να υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες ανασταλτικού χαρακτήρα μόνο για τα... όταν ζητείται η παρουσίαση των δεδομένων για τα ευαίσθητα, των δεδομένων. Υπάρχουν κάποιε πολιτικέ ομάδε οι οποίε ζητούν να υπάρχει κοινοποίηση ή δυνατότητα αναστολή μόνο όταν το πρόσωπο που ερευνάται βρίσκεται σε άλλο κράτο μέλο. Ή, αυτό επίση μπορεί να το πει εάν τα δεδομένα βρίσκονται σε άλλο κράτο μέλο από την εγκατάσταση του προσώπου. Θα επανέλθω. Μπροστά σε όλε αυτέ τι διαφορετικέ απόψει, ζήτησα από του συναδέλφου να κάνουμε μια συνάντηση των σκιωδών αρχή του μήνα και ζητήσαμε και την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και έναν δικαστή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και στη συνάντηση αυτή η νομική μας υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι η δική μου προσέγγιση στο προσχέδιο είναι νομικά ορθή. Επίσης επεσήμανε ότι η πρόταση ορισμένων πολιτικών ομάδων να πάρουμε τις διατάξεις από την οδηγία και πιο συγκεκριμένα αυτό που λέγεται να, ε, η πρόταση τους για το τι θα συμβαίνει σε περίπτωση που δεν υπάρχει νομική εκπροσώπηση του παρόχου στην Ευρώπη μας επιβεβαίωσαν ότι αυτό μπορεί να γίνει από νομικής απόψεως, ότι καλύπτεται από το άρθρο 82. Επίσης, ο δικαστής μας ξεκαθάρισε ότι οι λεγόμενες μόνο εθνικές υποθέσεις μπορεί να είναι μεν τέτοιες, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές αλλά και ο πάροχος δεσμεύονται από το δίκαιο που ισχύει στο κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένε ή διαμένουν. Επομένως δεν είναι τόσο απλό κανείς να παραμερίσει την αρχή της εδαφικότητας στην εφαρμογή του δικαίου. Επίσης, ακούσαμε ότι πολλές πολιτικές ομάδες ζητούν να είναι διαχειρίσιμο και ευέλικτο το σύστημα των κοινοποιήσεων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα, κάν, θα οργανώσουμε και άλλες συναντήσεις σκιωδών και τεχνικέ συναντήσει, ξεκινώντα από την επόμενη εβδομάδα, για να βρεθούν συμβιβαστικέ λύσει, ελπίζοντα ότι θα μπορέσουμε να πάμε σε ψηφοφορία το Μάρτιο. Δεδομένου ότι όλοι επιθυμούμε να καταλήξουμε σε ένα νομοθέτημα το οποίο να είναι ορθό από την νομική άποψη αλλά και πρακτικά εφαρμόσιμο, το οποίο να εξασφαλίζει τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων Είμαι σίγουρη ότι αν προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς, θα βρούμε μια λύση την οποία τελικά να μπορούν να υποστηρίξει μια ευρεία πλειοψηφία. Γνωρίζω ότι το θέμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας εργαστούμε λοιπόν όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά του Κοινοβουλίου και βεβαίω ε, καλώς ορίζουμε και την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των ε, διαθεσμικών διαπραγματεύσεων να μας εκθέσει τις απόψεις τη και πιο συγκεκριμένα αυτό που μας πρότεινε αν μπορεί να μας κάνει μια παρουσίαση για, τα για το τους ασφαλείς διάβλους ανταλλαγής στοιχείων θα ήταν πολύ χρήσιμο. Αναμένουμε λοιπόν κυρία Σίπελ την ε, ε, εξέλιξη αυτή την επόμενη εβδομάδα να ακούσουμε και τη δυνατότητα να υπάρξει ψηφοφορία το Μάρτιο. Αυτό θα ήταν πολύ καλή είδηση, δεδομένου του ότι αυτή η, αυτός ο είναι προφανώς πολύ σημαντικό και προκαλεί και μεγάλες διαστάσεις. Είναι πολύ διαφλονικούμενο. Όλοι λοιπόν... Θέλουμε να υπενθυμίσουμε πόσο απαραίτητο είναι να υπάρξει νομική βάση σωστή και ασφαλή σε ό,τι αφορά το άρθρο 82, ε, το οποίο προτάθηκε και εγκρίθηκε ως ε, νομική βάση από την νομική υπηρεσία. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση των ε, συμβιβασμών. Τώρα, να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, λέει ο Πρόεδρος. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε καθυστερήσει εξ αρχής. Και καταλαβαίνω βέβαια γιατί. Γιατί προσπαθούμε προφανώς να συμπτύξουμε τρεις ε, συζητήσεις στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διατάξης για τις επιστροφές και τις επανεισδοχές και γι' αυτό έχουμε μείνει πίσω. Να ακούσουμε τώρα τους εμπειρογνώμονες μας για το θέμα των ναρκωτικών. Έγινε λοιπόν μια αποστολή της Επιτροπής μας στην Λισαβόνα το 2019 και μας είπε ο επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας, η Κατερίνα Κινίτσι, η συνάδελφός μας, ε, στις αρχές του χρόνου, τι έγινε. Μας ε, είπε λοιπόν ειδήσει ανησυχητικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μετατρέπεται σε μεγάλο εργοστάσιο ναρκωτικών, για την εισαγωγή ναρκωτικών αλλά και για την παραγωγή ναρκωτικών. Έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό με τους πανελίστες μας. Έχουμε να καλωσορίσουμε και τον κύριο Αλέξης Γκουστέιλα από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά. Καλώς ορίσατε στη Λισαβόνα. Και τον κύριο Βιλ Φαν ο οποίος είναι από τη Γυροπόλα. Να ακούσουμε τις παρουσιάσεις τους και μετά θα ξεκινήσει γύρω ερωτήσεων και συζητήσεων με τους συντονιστέ. Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι έχουμε και την ψηφοφορία μπροστά μας. Μέχρι τις 11.45 η αίθουσα θα γεμίσει. Θα έρθουν ε, οι συνάδελφοι για να ψηφίσουν. Μπορούμε να βάλουμε την ψηφοφορία στις 12 το αργότερο. Ε, ένα λεπτό είναι η ψηφοφορία μια έκθεση Βόλαφ, τη συναδέλφου κ. Βόλαφ. Δεν θα πάρει πολύ ώρα λοιπόν η ψηφοφορία, αλλά να μην ξεπεράσουμε τις 12 η ώρα, γιατί δεν έχει νόημα να περιμένουν οι συνάδελφοι που έχουν έρθει για την ψηφοφορία. Το λόγο έχει λοιπόν ο κύριος Χόσδελ. Σας ευχαριστώ πολύ και ανυπομονούμε να ακούσουμε την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Μεγάλη μου χαρά που είμαι και πάλι εδώ στην Επιτροπή σας να σας παρουσιάσω τα βασικά πορίσματα σε ό,τι αφορά τη σκηνή έκθεση την οποία ε, με τη Europol και να ευχαριστήσω με τον συνάδελφό μου εδώ και όλους τους συναδέλφους της Europol. Σκοπός της έκθεσης αυτής είναι να γίνει μια στρατηγική ανάλυση με συγκεκριμένες στρατηγικές συστάσεις. Κάθε τρία χρόνια γίνεται η έκθεση αυτή. να δούμε τις διαφάνειες. Το πρώτο θέμα, λοιπόν, ότι το φαινόμενο των ναρκωτικών ε, κατίσταται πιο πολύ παραποτέ παγκόσμιο και ψηφιοποιημένο. Και λεπτομέρειες θα βρείτε στην έκθεση. Δεύτερο βασικό στοιχείο, ότι αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ναρκωτικών παρά ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ένα μήνυμα θέλουμε να σας μεταφέρουμε σήμερα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίκτυπος στην ε, πολιτική. Ποτέ δεν είχαμε τόσο πιο πολλά ναρκωτικά ε, διαθέσιμα, ε, συνθετικά ή φυσικά και με μεγάλη σε γνήσια μορφή. Πιο φθηνά παρά ποτέ κάτι επίσης καινούριο, το οποίο δεν ε, υπήρχε πριν από πέντε χρόνια σε αυτή τη διάσταση, είναι η αυξημένη βία και θέματα διαφθοράς σε σχέση με τα ναρκωτικά. Να σας υπενθυμίσω ότι πέρσι στην Ολλανδία δολοφονήθηκε ένας δικηγόρος. Σε κάποια κρατημέλη οι διαμάχες μεταξύ των συμμοριών γίνεται με χειροβομβίτες, με βόμβες, επιθέσεις φαινόμενα τα οποία στο παρελθόν τα είχαμε στο μυαλό μας για την Κεντρική Αμερική. Τώρα λοιπόν αυτά καταφθάνουν και συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου και η Ένωση και τα μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό επίσης είναι σημαντικό, γιατί ω τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε αυτό που ονομάζουμε την ισορροπημένη προσέγγιση των ε, ναρκωτικών, δηλαδή σε ό,τι αφορά επενδύσεις στην δημόσια υγεία και ε, δράσεις για την μείωση της διαθεσιμότητας. Σήμερα αυτό το μοντέλο αμφισβητείται. Το γεγονός είναι ότι οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και η βία αυξάνονται. Θα πρέπει να προσέχουμε λοιπόν και να δούμε τι μοντέλο μπορεί να εγγυηθεί τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία και προφανώ θα συνάδει και με τι αρχέ και τι αξίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να, δώσω δύο, να πω δύο λόγια για τον αντίκτυπο και για τι κινητήριε δυνάμει. Παρουσιάζουμε στην έκθεση μια συνολική προσέγγιση και μια συστημική προσέγγιση. Καταρχά, με λεπτομέρειε σε σχέση με τι κινητήριε δυνάμει τη αγορά ε, των ναρκωτικών, αλλά και τι συνέπειε. Ο συνάδελφό μου, ο Βίμ, θα σα παρουσιάσει ε, κάποια βασικά ζητήματα αναφορικά με το θέμα αυτό. Εδώ θα ήθελα να επιμείνω στο εξή. Αν μπορούμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια, ο χρηματοοικονομικό αντικτύπο των αγορών ναρκωτικών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υπολογίσουμε την έκταση της ε, αγοράς ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινήσαμε από τα δεδομένα που είχαμε σε ό,τι αφορά τη χρήση ουσιών και ναρκωτικών. Ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα ποσοστό χαμηλότερο του πραγματικού, αλλά τουλάχιστον βασίζεται στα μοναδικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία συνέλεξε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και τα σχετικά σημεία εστίασης. 30 δις λοιπόν υπολογίζονται. 30 δις ανά έτος σε επίπεδο λιανικής πώληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζεστε τώρα ότι τα χρήματα αυτά αυτά τα έσοδα από τα ναρκωτικά επανεπενδύονται σε σημαντικές και σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες. Και που και που φυσικά υπάρχουν και σχετικές ε, τρομοκρατικές ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα έσοδα αυτά. Ο αντίκτυπο τώρα τη αγορά ναρκωτικών, όπω παρουσιάζεται στην έκθεση, καταρχά σχέσει με τρομοκρατία και άλλε εγκληματικέ δραστηριότητε. Επίσης, έχουμε μια επιπρόσθετη ανάλυση και έρευνα για το σκέλος αυτό. Έχουμε τη βλάβη και τη ζημία προφανώς για τα άτομα, τις οικογένειές τους, τις κοινότητές τους, τις συνέπειες για την νόμιμη οικονομία και τέλος την διαφθορά και την επιβάρυνση των δημοσίων α, θεσμικών οργάνων. Όταν μιλάμε για πιο στρατηγική ανάλυση για το πώς έχει κατάσταση στην Ευρώπη, να επισημάνω το εξή. Η επιβάρυνση για το κράτος δικαίου και πόσο σημαντικό είναι το, η συνέπειε για τα άτομα. Ο, αυτά είναι φαινόμενα τα οποία έχουν επιτανθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Τώρα, να δούμε τις ομάδες των ουσιών, καταρχάς για την κάναβη και τα καναβοειδή. Εξακολουθεί να αποτελεί αυτή τη μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε μεγάλη καινοτομία στην αγορά και μεγάλη ποικιλομορφία των προϊόντων. Για όσους ήσασταν εδώ πριν από δύο χρόνια, να σας θυμίσω ότι πριν από δύο έτη σας ενημέρωσα την, για την κατάσταση και σας είχα πει για νέα προϊόντα τα οποία παράγονται στη ΣΥΠΑ γιατί πλέον υπάρχει και νόμιμη χρήση για αναψυχή των ναρκωτικών αυτών και σας είχα πει ότι σύντομα θα έχουμε την άφηξη των προϊόντων αυτών μέσω παράνομων οδών προφανώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφάτως λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε βρει ε, κάποιες ε, κάποια στοιχεία για άθμισμα προϊόντα τα οποία παράγονται στη ΣΥΠΑ και περιέχουν 70 έως 95% κάνα Άρα ο κίνδυνος, όπως σας είπα, είναι και παγκόσμιος και ψηφιοποιημένος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και να προετοιμαστούμε. Θα πρέπει επίσης ε, όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής στην εισαγωγή του, να λάβουμε υπόψη ότι η Ευρώπη έχει γίνει μεγάλος παραγωγός φυτικής κάναβης. Να αντιληφθούμε και τον κίνδυνο στην υγεία και τον ε, αντίκτυπο στο περιβάλλον που προκαλείται από την παραγωγή αυτή. Και αυτές οι περιβαλλοντικές απειλές προφανώς μπορούν να συνδεθούν και ακόμα περισσότερο με την παραγωγή νέων συμφετικών και ψυχοτρόπων ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ηρωίνη και άλλα οπιοειδή εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά φυσικά την υγεία και το κοινωνικό κόστος. Έχουμε νέες εξελίξεις στην παραγωγή ροήνης και αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση και τον ε, έλεγχο χημικών ουσιών πρόδρομων. Και έχουμε φυσικά και προβλήματα σε ό,τι αφορά την νότια διοδό, το κανάλι του ΣΟΕΣ συγκεκριμένα, του Για την επιτροπή σας έχω να πω το εξή ότι δεν μπορούμε να ε, αποσυνδέσουμε αυτά τα κανάλια, αυτές τις διόδους ε, προμήθειας, ιδιαίτερα από την Ασία, με τις νέες εμπορικές οδούς. Για παράδειγμα, μα, τους δρόμους του μεταξιού που προωθούνται από την Κίνα και τον αριθμό των λιμανιών. Που αποτελεί κινέζικη αρμοδιότητα. Εδώ τονίζεται λοιπόν η ανάγκη για στενήτερη συνεργασία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά του ελεγχού. Σε ό,τι αφορά την κοκαίνη τώρα. Θα δείτε, θα έχετε ακούσει κάποιοι από εσά ότι προσφάτω υπάρχει τεράστια αύξηση και μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά τι οδού τράφικινγκ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το λιμάνι του Ρότερνταμ που έχει μεταφερθεί στο λιμάνι της Αμβέρσας. Πριν από ένα χρόνο, δεν κάνω λάθος, είχαμε 50 τόνους κοκαίνη που κατασχέθηκαν στην Αμβέρσα και μόνο. Και άλλοι 50 τόνοι οι οποίοι εντοπίστηκαν με τελικό προορισμό πάλι το λιμάνι της Αμβέρσας. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αύξηση και στις κατασχέσεις παντού. Πριν από τέσσερα χρόνια ήταν σαφές ότι η κατάσχεση πάνω από το 50% της ε, κοκαίνης που έφτανε στην ε, Ευρώπη μέσω του ΑΜΦ του τώρα αυτό το ρόλο το παίζει το λιμάνι της Αμέρσας. Και η Βόρειος Αφρική συχνά είναι η περιοχή διέλευσης, κυρίως σε ό,τι αφορά το Μαρόκο, κυρίως επειδή ε, έχουμε παράνομες οργανώσεις, ε, συμμορίες στην, ε, στο Βελγίο και στην Ολλανδία που χρησιμοποιούν το Μαρόκο ε, ως κόμβο πρωτού καταφτάσουν τα προϊόντα αυτά στην Ευρώπη. Κάτι άλλο τώρα για ένα άλλο θέμα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συνέπειες της χρήσης κοκαίνης. Βλέπουμε μεγαλύτερη, τεράστια αύξηση της διαθεσιμότητας κοκαίνης. Και αυτό μπορεί να μην φαίνεται στα τυποποιημένα προγράμματα απεξάρτησης αυτό όμω που διαπιστώνουμε σε πολλέ πόλεις και στι Βρυξέλλες μεταξύ αυτών είναι η αύξηση τη χρήση κοκαίνης κράκ, το οποίο παλιά τα τελευταία 20 χρόνια περιοριζόταν σε κάποιες λίγε πόλεις. Άρα, αν δεν βλέπουμε ποσοστιαία αύξηση της κατανάλωση ακόμα, αυτό ακόμα δεν έχει εντοπιστεί φυσικά στο ραντάρ, αν και τα πρώτα στοιχεία έρχονται για την αλλαγή Τη στοιχείου αυτού είναι ότι δεν χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιούταν η κοκαίνη. Χρησιμοποιείται πλέον σε μορφή κρακ κοκαίνης που έχει πιο σοβαρές συνέπειες για την δημόσια υγεία. Για τις αμφεταμίνες και τις μεταμφεταμίνες, MDMA, εδώ κοιτάζουμε πόσα σημεία παραγωγής έχουμε πλέον, μεγάλη εξάπλωση σε σχέση με το 2015 έως το 2017. Οι συνάδελφοι από την Europol θα έχουν περισσότερα στοιχεία επιχειρησιακά και λεπτομέρειες, αλλά βλέπετε πόσα πολλά σημεία παραγωγής, πόσο επεκτάθηκε η παραγωγή. Ξεπερνά και τα γνωστά σημεία παραγωγής πριν από 10-15 χρόνια κατά πολύ. Πάντω ε, την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε με μερικού Αμερικανούς συναδέλφου και πραγματικά μας ανησυχεί η πληροφορία ότι υπήρχε μια μεγάλη μονάδα παραγωγής μεταμφιμινών στην Ολλανδία που λειτουργούσε χάρη στην υποστήριξη και μεξικανικών καρτέλ. Και κάτι που θα μας αποσχολήσει στο μέλλον και θα χρειαστεί ευρωπαϊκή συντονισμένη δράση είναι ότι οι διασυνοριακές ομάδες ε, οργανωμένου εγκλήματος θα θεωρούν, θεωρούν ήδη την Ευρώπη ως ένα από τα πεδία που μπορούν να δράσουν ανενόχλητοι. Τώρα για τις νέες ψυχοτρόπες ε, ουσίες, βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια ότι οι έντονες κουκίδες είναι οι νέες ουσίες που έχουν ε, βρεθεί και εντοπιστεί στην ε, Ευρωπαϊκή Αγορά το 2018, ήδη σήμερα, Μπορώ να σα δώσω κάποιε πρόσφατε πληροφορίε. Ο συνολικό αριθμό τέτοιων ουσιών που έχουμε παρατηρήσει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 780. Θα ήθελα τώρα να φτάσω σε συμπεράσματα για να εξοικονομήσουμε κάποιο χρόνο για τη συζήτηση είναι η στιγμή πραγματικά να ξυπνήσουμε και να αντικρίσουμε την πραγματικότητα και να δούμε κάποιες σαφείς συστάσεις ως προς τη χάραξη πολιτικής, διότι οι πληροφορίες αυτές έρχονται ακριβώς τη συγκυρία όπου το Συμβούλιο και η Επιτροπή μαζί με το Κοινοβούλιο θα συζητήσουν την αξιολόγηση της ε, τρέχουσας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενδεχόμενη οθέτηση μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγικής, ώστε να υπάρχει μια σφαιρική προσέγγιση. Αυτό που σα έδειξαν αυτά τα δεδομένα και νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό μήνυμα τη διευθύντρια τη Europol και το δικό μου, τη κυρία Δεμπολ, όταν ε, ετοιμάσαμε την έκθεση αυτή, είναι ότι πρέπει να συνέλθουμε και να ξυπνήσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ναρκωτικά να μην αναφέρονται καν στις 10 πρώτε προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν συναντώνται Υπουργοί Ιστορικών, α πούμε. Ε, είναι πραγματικά μια πυρολογιακή βόμβα. Θα πρέπει να την ε, απενεργοποιήσουμε και πρέπει επιτέλους να περάσουμε στην δράση. Ακόμα και στο πλαίσιο της συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να αποδώσουμε στα ναρκωτικά την προσοχή που τους αναλογεί. Είναι σοβαρότατες απειλές και για την εσωτερική ασφάλεια Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι χάρη σε ή εξαιτία των δράσεων του συνόλου δράσεων που ανέπτυξαν τα κάτι μέλη για να αντιμετωπίσουν την επιδημία εντό αγωγικών ερωίνης πριν από 20 χρόνια, κάτι καταφέραμε. Τώρα έχει συμβεί το ανάποδο σε σχέση με την αντιμετώπιση των νέων ουσιών. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να περιμένουμε να έχουμε πάλι ένα φαινόμενο όπως στις ΗΠΑ επιδημία, επιδημίας. Να θυμίσω ότι είχαμε 72.000 θανάτους πριν από δύο χρόνια ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες από θανάτου λόγω κατανάλωσης οπιοειδών. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, αλλά υπάρχει τέτοια προσφορά στην αγορά, τέτοια διαφορία για, την, ε, για τον περιορισμό ζήτηση για τα ναρκωτικά, που αν νομίζουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα έχουμε ήδη χάσει πάρα πολύ χρόνο για να αντιμετωπίσουμε μια νέα επιδημία. Έχουμε λοιπόν τώρα τη δυνατότητα, έχουμε του πόρου να συνεργαστούμε και με το δικό μα τον οργανισμό και με τη Europol και με το δίκτυο και με του διαφορού ε, συνεργάτε μα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανεί. Εάν δεν υπάρξει η κατανόηση του φαινομένου σήμερα, θα είναι πολύ λίγα για δράση σε λίγο. Και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι έχουν γίνει ως τώρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοστέλ. Εγώ θα έλεγα η παρουσίαση του εκτελεστικού διευθυντή της Europol να είναι πολύ συντομότερη, διότι έχουμε 12 παρα 10 ψηφοφορίες. Θα είναι μεν σύντομη ψηφοφορία, αλλά δεν μπορούμε να την αναβάλουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ ε, σύντομα για να μπορέσουμε να ακούσουμε τα σχόλια και των συναδέλφων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ και σε συνεργασία με τον MCDA για να παρουσιάσουμε το πλαίσιο συνεργασία των δύο οργανισμών. Οι εξελίξεις που παρουσίασε ο Αλέξη ε, κατά το κάνουν σαφέ. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τους διεθνεί οδούς εμπορία είναι σοβαρή προτεραιότητα και της Europol και των διοκτικών αρχών. Έχουμε διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα σε ευρωπαϊκές αγορές. Σας δόθηκαν πολλά παραδείγματα. Τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι πρέπει να επιτείνουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε το διασυνοριακό έγκλημα, δίνοντας αυτό το φαινόμενο ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζονται όμως περισσότερες προσπάθειες. Στη διαφάνεια αναφέρθηκε από τον Αλέξη. Βλέπετε ποια είναι η προσέγγισή μας. Μα μίλησε για, το για τους λόγους που προκαλούν τα φαινόμενα αυτά, την αποκοσμοποίηση, πώ διοργανώνται οι διασυνορικές ομάδε εγκλήματο, πώς αξιοποιούν τα τεχνολογικά μέσα και τι μπορούν να κάνουν οι διοκτικές αρχές και οι διάφοροι φορείς για να απαντήσουν σε όλα αυτά. Επόμενη διαφάνεια αντίκτυπος, επιπτώσεις στην κοινωνία, στην αγορά ναρκωτικών. Εγώ να ε, πω περισσότερα λίγο για την εξέλιξη του οργανωμένου κλίματος και τι σημαίνει για αποτελεσματική απόκριση των διοκτικών αρχών. Θα αναφέρω κάποιες χώρες, αλλά είναι σαφές όπως τόνισε και ο Αλέξης, ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό, διεθνές. Δεν αφορά μόνο ορισμένε χώρες. Επόμενη διαφάνεια. Να ξεκινήσω με τα βασικά μηνύματα που εντοπίσαμε και στην έκθεσή μας από την πλευρά των διοκτικών αρχών. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τονίσω το οργανωμένο έγκλημα είναι κατά την άποψή μας ο πιο η πιο σημαντική απειλή κατά την ασφάλεια των ε, κρατών μελών. Η ενδιάμεση αναθεώρηση ΣΟΚΤΑ δείχνει ότι η δράση των οργανωμένων ε, ομάδων γίνεται περιπλοκότερη πολύ ε, περισσότερο διασυνοριακή και εμπλέκονται και φορεί και πολλέ φορέ και κυβερνήσεις. Το βλέπετε και στην έκθεση. Το να αντιμετωπίσουμε τα νοικοτικά σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα και είναι σοβαρότατο η πηγή εισοδήματο για το οργανωμένο έγκλημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διεθνή αγορά τα νοικοτικά. Για να δείτε εδώ τι εξελίξει, δείτε δύο εικόνε επιχειρήσει που υποστηρίξαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό ήταν πριν από 10 χρόνια στην Ολλανδία. Εκείνη τη στιγμή ήταν η πιο προηγμένη μονάδα παραγωγής. Αλλά μετά περνάμε στο 2020 και έχουμε φτάσει εδώ. Βλέπετε από την εικόνα και μόνο ότι έχουμε φτάσει σε βιομηχανικά επίπεδα. Παράγονται πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Εξού και ο κίνδυνος για την κοινωνία μας. Αλλά πέρα από τα συνθετικά ναρκωτικά, μπορεί κανείς να φέρει εδώ αριθμητικά στοιχεία για να το υποστηρίξει όπω είπε και ο Αλέξ. Όμω στην Ολλανδία το τελικό αποτέλεσμα Ε, το ποσό, το κέρδος συνολικά ήταν 19 δις ε, ευρώ μόνο από τα συνθετικά ναρκωτικά στην Ολλανδία. Για τους συγκεκριμένους αριθμούς τώρα. Κέρδος που μπορούν ε, να εισπράξουν οι οργανωμένες ομάδες και οργανωμένες επιχειρήσεις που πράγουν την διαφθορά. Πίσω στη διαφάνεια τώρα. Το οργανωμένο έγκλημα η διακίνηση που εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών είναι το πιο ισχυρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και με τα πυροβόλα όπλα, με την πειρατεία, με τη διαφθορά, με την ε, ε, εμπορία παράνομων αποβλήτων. Σε όλα αυτά μπλέκονται οι ίδιοι. Επίση, για το πώ διορθώνονται, μπορούν να ελέγξουν όλη την αλυσίδα ε, πώληση κοκαίνης από τη στιγμή της παραγωγής μέχρι την, το σημείο πώληση και με έσοδα σε όλη την Ευρώπη. Έλεγχο ασκούν και στις αγορές της Ευρώπης αλλά και στις χώρες παραγωγής στη Λατινική Αμερική. Οι ομάδες αυτές είναι οργανωμένες ε, με το είδος με, το, με τη λογική της μαφίας. Δεν είναι μόνο την Ιταλική μαφία, ενώ τη μαφία που έχει προεκτάσεις και απλοκάμια διεθνώς είναι πολλέ οι μορφέ εγκλήματο που μπορούν ε, να οργανώσουν ταυτόχρονα. Είναι και άλλε οι οργανωμένε ε, ομάδε που εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν όλο ένα και μεγαλύτερε επιπτώσει. Ξέρουμε του Κολομβιανού, του Χιλιανού, του Μεξικανού με του ε, Κινέζου, του Νιγηριανού. Είναι οργανωμένε ομάδε που έχουν πλοκάμια και στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και τι περισσότερε φορέ οι δραστηριότητε των οργανωμένων αυτών ε, ομάδων έχουν ε, σχέση και με το εμπόριο ναρκωτικών, με τη διακίνηση ναρκωτικών. Σε σχόλια όπω η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, έχουμε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Το 2019 στη Σουηδία, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε 354 περιβολισμού και 30, 30 θανάτους ή τραυματισμούς Όλα αυτά σε σχέση με την αγορά ναρκωτικών, την αγοραπολισία ναρκωτικών. Επίσης με τη διαφθορά οι οργανωμένες ομάδες μπορούν να ε, δυσδύσουν σε πολιτικούς φορείς και οργανισμούς, προκαλώντας και άλλα φαινόμενα. Για να σας πω, ας πούμε ένα παράδειγμα, 250.000 ευρώ μπορεί να πάρει ένας τελωνιακό υπάλληλο για να κάνετε στραβά μάτια σε ένα φορτίο ναρκωτικών και επίσης για την ε, λεύκανση προσόδων μπορεί να δώσουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά αυτές οι οργανωμένες ε, ομάδες. Επίσης οι τεχνολογικέ λύσεις και καινοτομία μπορούν να βοηθήσουν την αγορά να γίνει παραγωγικότερη. Στο διαδίκτυο μπορούν να βρουν νέου πελάτες και να αυξήσουν το πελατολογιό τους. Δύο τρίτα είναι το σύνολο των ε, ερευνών που έχουν σχέση με ηλεκτρονικό ε, εμπόριο ναρκωτικών. Και εδώ ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα ευρωπαϊκά κράτη, να τα υποστηρίξουμε, να ελέγχουν τη δράση στον κυβερνοχώρο με όποια κίνηση μπορούν. Για το νομικό πλαίσιο επίκειται η συζήτηση, αλλά η τεχνολογία προσφέρει πολύ σημαντικά εργαλεία με την κωδικοποίηση ε, γιατί για να αποκρυπτογραφήσουν τα στοιχεία αρχές ε, έχουν φοβερέ δυσκολίες στις περισσότερες ε, υποθέσεις. Εδώ λοιπόν θα χρειαστεί μια νέα πρόταση με την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τελευταίο, ε, επίση σημαντικό, βλέπουμε την ανάδυση νέων γεωγραφικών περιοχών που γίνονται κόμβος και hub για την ανάπτυξη, γίνονται αιστεία παράνομων δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω για την εμπορία ναρκωτικών. Βλέπετε βέβαια πόσο σημαντική είναι η Λατινική Αμερική ούτω ή άλλω, αλλά έχουν πάρει μεγάλη αξία και τα Βαλκάνια. 60% τη κοκαίνης που παράγεται στην Κολομβία προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά και το 90% όλων των φορτίων κοκαίνης από τη Βραζιλία πάλι στην Ευρώπη πηγαίνουν. Οπότε να πάω στις ε, πιθανές απαντήσεις στο ποιε είναι οι επιπτώσεις για τις διοικητικές αρχές. Για να επανέλθω στις αρχικές μου παρατηρήσεις, υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη στις έρευνές τους, διότι μιλάμε για έρευνες με μεγάλη, ε, με πολλές απαιτήσει που είναι απαιτούν την υποστήριξη των ιδιωτικών αρχών, κάτι που κάνουμε από το 2018 συστηματικά. Πρέπει και τα, τις μεμονωμένες περιπτώσεις και τις ε, οργανωμένες ομάδες, να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού και να έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχημένη κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από το οργανωμένο έγκλημα και την ε, εμπορία ναρκωτικών. Και από το 2018 είχαμε τουλάχιστον 24 ομάδες κρούσης με 49 ε, στόχους προτεραιότητας και θεωρούμε ότι με τις κατασχέσεις μας πετύχαμε να ανακτήσουμε 84 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας γεωγραφικά και επιχειρησιακά και να δώσουμε έμφαση σε περιοχέ όπου υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και να εντείνουμε τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών τα καρτέλ των Βαλκανίων, ας πούμε, σας είπα ότι συνεργάζονται και με άλλες ομάδες της ΕΠΑ. Θα πρέπει όμως να σπάσει αυτή η αλυσίδα για να μην έρχονται και άλλα νοικοτικά στην Ευρώπη και επίσης πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογία. Έχουμε πει ότι η επικοινωνία, τα κρυπτονομίσματα, η κρυπτογράφηση είναι προκλήσεις για τις διοκτικές αρχές της Ευρώπης. Για το 2020 ένας βασικός στόχος είναι να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε τους φορείς, ε, τους αστυνομικούς, τις διοκτικές αρχές στο μέτωπο αυτό. Επίσης θα πρέπει να ενδυναμωθεί η ε, εντολή για την κατάσχεση ε, εσόδων από το οργανωμένο έγκλημα. Για την ώρα έχουμε μόνο 5% επιτυχία σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, κάποιοι αναφέρουν και τον αριθμό του, 1, του 1%. Πρέπει λοιπόν να τα πάμε καλύτερα και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η φυστάμενη νομοθεσία μεταξύ των 100 μελών θα ενερμονιστεί για να έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε για την λεύκανση, για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του σοβαρού εγκλήματος και το ξέπλυμα. Εδώ λοιπόν να πω πώς σκοπεύουμε να χαράξουμε τη στρατηγική μας όχι μόνο από την πλευρά των διοκτικών αρχών και της Europol, αλλά και το τι θα πρέπει να κάνουν και οι πολιτικοί θενούντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας Και υπάρχει και υψηλό κίνδυνο με τι πλατφόρμε του οργανωμένου εγκλήματο. Ε, ανέφερα το τελευταίο. Αν δείτε τι κούρσα υπάρχει για την παραγωγή των συνθετικών ναρκωτικών, από το 2015 και μόνο υπήρχαν ε, μόνο 900 και μόνο υπήρχαν 900 περιπτώσεις παράνομων αποβλήτων που περιβαλλοντικά βαρύνουν ε, το, επιβαρύνουν το περιβάλλον και τις κοινωνίες. Και τέλος πάντων μια έκκληση για δράση εδώ εν τέλει, γιατί ανυπομονούμε να συνεργαστούμε και μαζί σας και με τους συναδέλφους μας για να υποστηρίξουμε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Όπως συνήθως θα δώσω το λόγο στους συντονιστές. Θα ήθελα να σας ζητήσω να απευθύνετε ερωτήματα ευθέως στους ομιλητές μας, γιατί υπάρχουν και άλλα μέλη της Επιτροπής που έχουν ζητήσει το λόγο. Βοηθήστε μας λοιπόν. Ξεκινώ με εσά κύριε Πίτερ, που εκπροσωπείτε το ΕΛΚ. Σα ευχαριστώ. Σύντομα, ευχαριστώ του ομιλητέ και το κέντρο για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση και σημαντική. Είπατε ότι εκτιμάται την αξία στη Λιανική περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ των ναρκωτικών και ότι αυτό θα πρέπει να μας σοκάρει και να θεωρήσουμε ότι είναι μεγάλη προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και για τα κρατημέλη. Δεύτερον είπατε ότι είναι αυτός ένας τομέας στον οποίο χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία, στενή συνεργασία των κρατών, τα ναρκωτικά. Δύο ερωτήσεις, παραγωγή κοκαίνης στη Νότια Αμερική και στην ηρωίνη στο Αφγανιστάν έχουν φτάσει το ιστορικό τους υψηλό. Ε, οι προσπάθειες μας για συνεργασία με τις χώρες αυτές έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς και το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο ζητήματα στην εξωτερική μας πολιτική. Δεύτερο ερώτημα, οι δράσεις των διοκτικών αρχών που σημείωσαν επιτυχίες κατά των διαφόρων ψηφιακών ε, χώρων αγοράς ναρκωτικών θα βασίζονται όλο και περισσότερο στις νέες τεχνολογίες για να έχουμε τις επιτυχίες. Επομένως, σας ρωτώ ποια μέτρα νομίζετε εσείς ότι χρειάζεται να υιοθετήσουμε γρήγορα και επίσης ποια είναι η δική σας αξιολόγηση του σημερινού συστήματος συνεργασίας. Ευχαριστώ. Κυρία Σίπελ, γρήγορα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα και στην αρχή, έγινε αποστολή στις υπηρεσίες αυτές, επομένως, και έχουμε και τη σχετική έκθεση, επομένως εγώ θα απευθύνω συγκεκριμένα ερωτήματα και παρατηρήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε πρόβλημα επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, καταναλώνουν, τους αρέσουν τα ναρκωτικά, είτε μιλάμε ε, οι εγουσίες που, στις οποίες μπορεί να εφιστεί κανείς, γιατί αυτό συμπεριλαμβάνει και το αλκοόλ, αλλά φτάνουμε μέχρι και τις παράνομες ε, αυτό δεν σημαίνει ότι προωθώ την νομιμοποίησή τους, αλλά υπάρχει ένα θεμελιώδες, αν θέλετε, πρόβλημα. Αναφερθήκατε στην κάναβη. Γνωρίζετε ότι για ορισμένους ανθρώπους η κάναβη ε, είναι χρήσιμη, τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν, για παράδειγμα, χρόνιο πόνο, σε ασθενείς με καρκίνο. Όμως, είπατε ότι μπορεί αυτό να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τι ακριβώς εννοείτε. Μετά, όσον αφορά τη χρήση ηρωίνης, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γνωρίζουν όλες οι χώρες ποιες είναι οι συνέπειες της αύξησης της χρήσης της. Γνωρίζω για παράδειγμα ότι στη Γερμανία ακόμα και σε ορισμένες περι, περιπτώσεις, έχουμε ορισμένε περιπτώσει, μάλλον σε περιοχέ τη χώρα, αύξηση της χρήσης ε, ηρωίνης. που την ανοιχνεύουμε με την ύπαρξη ριών στο νερό. Ε, έχετε αναλάβει ε, κάποιες δράσεις για να ευαισθητοποιήσετε τις τοπικές αρχές. Είπατε ότι όλοι και περισσότερο χρησιμοποιούν πια αυτά τα κυκλώματα τα και ε, εμπορευματοκιβώτια και συγκεκριμένους τρόπους διακίνησης. Τι σημαίνει αυτό για τους συνοριακούς ελέγχους, τι θα πρέπει να αλλάξει στον έλεγχο των κοντέινερ και σε σχέση με τα συνθετικά ναρκωτικά. Διαπιστώνουμε ότι πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλος παραγωγός συνθετικών ναρκωτικών. Τι χρειάζεστε για να εντοπίσετε πού παράγονται αυτά τα συνθετικά ναρκωτικά και τι είδους περισσότερη βοήθεια θα μπορούσαμε να σας προσφέρουμε για να είστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτό. Κύριε Εντφέλτ, δεν θέλετε. Το λόγο ευχαριστώ. Ε, Κυρία Παγασουτούντα, είχατε ζητήσει το λόγο σύντομα. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, της χώρας μας διαπιστώσαμε νέοι να συμμετέχουν σε οργανωμένες ομάδες εγκληματικές που να συμπεριφέρονται σαν να ήταν ήρωες της σειρά Νάρκος, την τηλεοπτική. Ο ε, διαπιστώνουμε αύξηση του αριθμού των θανάτων εξαιτίας ναρκωτικών. Ε, χρήσιμο θα ήταν να μου το επιβεβαιώσετε αυτό αν μπορείτε να μου δώσετε κάποια αριθμητικά στοιχεία και για την Ευρώπη και για άλλες περιοχές του κόσμου. Ε, επίσης γνωρίζουμε ότι η χρήση οδηγεί σε ψυχιατρικά ε, προβλήματα, προβλήματα ψυχικής υγείας. Και αυτή, αυτό το ζήτημα συχνά το αφήνουμε στην άκρη γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς πρέπει να το λύσουμε ή προσπαθούν να το κρύψουν οι οικογένειες. Τι κάνουμε γι' αυτό. Μετά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να γνωρίσει καλύτερα η κοινή γνώμη ποιες είναι οι ουσίες αυτές οι οποίες είναι πιο επικίνδυνες και πιο θανατηφόρες. Για τους πράσινους, η κυρία Μπρικμό. σας ευχαριστώ, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και χαίρομαι όταν ακούω κάποιου ε, ανθρώπου να μιλούν για τέτοια θέματα χωρί να ακολουθούν, να ακολουθούν ξύλινη γλώσσα. Ε, το, η κατάσταση στο λιμάνι της Αμβέρσας που αναφέρατε είναι πολύ ανησυχητική και έχει δημιουργήσει και προβλήματα στην περιοχή, ε, κοινωνικά προβλήματα, βία στην περιοχή αυτή, το αναφέρατε κι εσείς. Μιλάμε ότι ορισμένοι, μαθαίνουμε ότι ορισμένοι μπορούν να κερδίζουν μέχρι και 5.000 ευρώ την εβδομάδα με αυτή τη διαφθορά, ότι έχουμε επίσης λιμενικούς οι οποίοι λαδώνονται για να κλείνουν τα μάτια στην Αμβέρσα. Ε, έχουμε επίσης ανήλικους να συμμετέχουν στις εγκληματικέ ομάδες, μέχρι και 14 ετών παιδιά έχουμε διαπιστώσει, με όλες τις μακροπρόθεσμες κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει αυτό και επίσης ότι ορισμένοι το χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν αυτή την κατάσταση για να ρίξουν λάδι στη φωτιά κάποιων εντάσεων σε κοινωνικό επίπεδο στην περιοχή, προσπαθώντας να στοχοποιήσουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Όλα αυτά διαπιστώνω στο λιμάνι. Ε, θα ήθελα να μου πείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα, δηλαδή για να αντιμετωπίσει ζητήματα ένταξη των νέων, ε, φροντίδα κοινωνική των νέων, τις, ε, να του ε, βοηθήσει να πάνε στο σχολείο, πέρα δηλαδή από την αστυνομική δίωξη των εγκλημάτων. Γιατί συχνά αυτό που ακούμε από εκείνου που εργάζονται στο πεδίο είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι και αύξηση των ελέγχων, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό λείπει στην Αμβέρσα, αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία. Ευχαριστώ. Υπάρχει εκπρόσωπο του ID. Κάποια ερώτηση. Όχι. ECR τότε. Ούτε από το ECR. Η Γκουέ θα ήθελε κάποιο το λόγο. Ναι, ε, παρακαλώ. Κύριε Αρβανίτη. Excuse me, Αβρανίτης. Αβρανίτης. Η παρουσίαση για άλλη μια φορά ήταν εξαιρετική και πάρα πολύ χρήσιμη για άλλους συναδέλφους. Όμως ε, πριν θέσω ένα μόνο ερώτημα θέλω να σημειώσω ένα πράγμα μόνο. Βασικό πράγμα που αφορά στην χρήση και στην εξάρτηση είναι η ανάγκη των ανθρώπων να κάνουν χρήση και να εξαρτώνται. Διότι μην πάμε σε μια λογική πολιτικής ή πολέμου ουσιών, διότι πολλοί χρήστες πίνουν κόλες, πίνουν βενζίνη, πίνουν πράγματα τα οποία είναι στην ομιμότητα. Οπότε είναι λάθος να μπούμε σε μια λογική νόμιμης και παράνομης ουσίας, αλλά πρέπει να δούμε τη βασική ε, αξία γιατί ένας άνθρωπος επιλέγει να πεθάνει. Ρωτώ, η ανάγκη λοιπόν είναι το βασικό ζήτημα και να δούμε. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη μιας ενιαίας πολιτικής στρατηγικής για τις χώρες μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βόμβα που περιγράψατε στην εισήγησή σας. Και ένα δεύτερο, Πρόεδρε Αλέξη, θα ήθελα να ρωτήσω πόσες νέες συνθετικές ουσίες παράγει η παράνομη βιομηχανία στην Ευρώπη, στον κόσμο, καθημερινά. Ευχαριστώ. Και τώρα δύο ακόμα συνάδελφοι και παρακαλώ σύντομα, διότι είναι σαφές ότι αρχίζει να γεμίζει ασφικτικά η αίθουσα λόγω της ψηφοφορίας. Πρώτα ο κύριος Λένας και μετά η κυρία Ίντζερ αν δεν κάνω λάθος. Και μετά πολύ γρήγορα και πάλι ο λόγος στους προσκεκλημένους μας για να απαντήσουν. Κύριε Λένερς, ευχαριστώ σας, ευχαριστώ και χαίρομαι πολύ που έρχονται τόσοι για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως τα ναρκωτικά στην Ευρώπη. Από την πλευρά της Ολλανδίας, διότι είμαι πάντοτε πολύ περήφανος, όταν η Ολλανδία είναι πρώτη στις ε, ταξινομήσεις διεθνώς, αλλά αυτό που δεν καταφέραμε με το ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια, το καταφέραμε με τα ναρκωτικά με τη μία, από ό,τι φαίνεται. Οι κάτω χώρε είναι 250 φορέ μέσα στην έκθεσή σα κάπου. Δεν μα κάνει να καμαρώνουμε φυσικά αυτό, διότι για την κάναβη και την κοκαίνη είμαστε από του μεγαλύτερου παραγωγού των συνθετικών. Ε, παράγουμε νέε ψυχοτρόπε ουσίε. Όλα αυτά είμαστε πρώτοι. Ευχαριστώ λοιπόν και τους δύο μιλητές που το υπογραμμίζουν. Είναι σημαντικό να τονίζονται όλα αυτά δεδομένη και της τωρινής συζήτησης που γίνεται στα πολιτικά αυτή τη στιγμή για το πώς μπορούμε όχι να αντιμετωπίσουμε την αγορά ναρκωτικών, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε την αγορά ναρκωτικών στην ε, Ολλανδία με κάποιες νομιμοποίησεις. Εσείς πώς θα βλέπατε μια τέτοια νέα πολιτική των κάτω χωρών εφόσον εφαρμοζόταν. Και αν δεν μπορείτε να σχολιάσετε συγκεκριμένε χώρε, εν γέννη, εάν ένα κάτω μέλο από τα 27 αποφασίσει να, να νομιμοποιήσει σκληρά νοικοτικά, τι θα σήμαινε αυτό από την ε, ευρωπαϊκή πρόπτικη, διασυνοριακά, τι θα συνέβαινε αν οι υπόλοιποι 26 συνέχιζαν να τα απαγορεύουν και να τα καταπολεμούν. Ε, και, τα ναρκωτικά και την καταναλωσή του και το οργανωμένο έγκλημα. Από την, από την ευρωπαϊκή λοιπόν πλευρά τι θα σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και για αυτή την πολύ σημαντική ενημέρωση. Ε, λέγεται ότι μια από τις σημαντικότερες ε, στρεβλώσεις της αγοράς ναρκωτικών είναι ότι οι νέοι ε, χάνουν τις ζωές τους. Οι νέοι ε, ακριβώς λόγω της συμμετοχή σε συμμορίες και οργανωμένες ομάδες με δολοφονίες χάνουν τη ζωή τους. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε πώς αναπτύσσεται ο αλληλοσχετισμός μεταξύ ε, ανθρωποκτονιών και δολοφονιών και της χρήσης ναρκωτικών ή της συμμετοχής σε οργανωμένες ε, ομάδες. 10 από 28 ε, κράτη-μέλη μόλις, ε, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, συλλέγουν συστηματικά στοιχεία για το θέμα αυτό. Ε, δεν είναι λοιπόν ε, συστηματική συλλογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μας απασχολεί πολύ. Πρέπει να βρούμε δραστικές λύσεις σε όλες τις χώρες αλλά και μεταξύ των χωρών σε συνεργασία. Τι θα κάνετε λοιπόν για τη συλλογή συγκρίσιμων στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια τελική ερώτηση όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, τι μέτρα μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι τα πιο σημαντικά για την καταπολέμηση των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. Μπορείτε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο για τις εταιρικές σχέσεις που αναφέρεται και στο κεφάλαιο επιχειρησιακές αποκρίσεις. Ευχαριστώ κύριε Έντφελτ. Ε, το χρονομιλία σας. Είπατε ότι θέλετε το λόγο. Ναι, 32 δεύτερα, γιατί θέλω να απαντήσω λίγο σε αυτά που είπε ο συνάδελφο ο κ. Λέιναρ σε ό,τι αφορά μια Ολλανδική συζήτηση. Ολλανδο-Ολλανδική συζήτηση που την έφερε στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα σχολιάσω το πόσο έκανε καρικατούρα το κόμμα μου, όσο και να σχολιάσω πόσο αποτυχημένος και Ακριβώ είναι αυτό ο πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Γιατί και εμεί ανησυχούμε για την υγεία των πολιτών και θέλουμε να δοθεί ένα τέρμα σε αυτή την ε, εγκληματικότητα και τη συμμορία πολέμου. Σε ό,τι αφορά το παράνομο dumping επίση ε, στη φύση τοξικών ουσιών. Αλλά έχουν αποτύχει όλα αυτά. Α προσπαθήσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλη μέθοδο. Ευχαριστώ πολύ και να ακούσουμε τώρα του πανελίστε μα. Αν θα μπορούσατε παρακαλώ να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ετέθησαν, να έχετε υπόψη σας στο χρονικό όριο ότι κανονικά έπρεπε να ψηφίζουμε τώρα. Μάλιστα, να απαντήσω κάποιες από τις ερωτήσεις σας και θα σας στείλω και κάποιο σημείωμα για να σας δώσω και σε διμερείς συναντήσεις, αν θέλετε, πιο λεπτο, λεπτομερείς πληροφορίες. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας καταρχάς και κάποιοι από εσάς διαβάσατε την έκθεση. Αυτό είναι εξαιρετικό για μας. Να ξεκινήσω από την ε, ερώτηση που έκανε ο κ. Πέτερς. Να πω ότι τμήμα της απάντησης θα δοθεί από λειτουργικής πλευράς, από τον συνάδελφο της Europol. Θα πρέπει να ενισχύσουμε, θεωρώ, τη συνεργασία αυτό σημαίνει να συνεχίσουμε να συλλέγουμε αποδεικτικά στοιχεία. Και ω εκ τούτου υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, όχι μόνο για την κοκαίνη, το ίδιο ισχύει και για την ηρωίνη και για άλλε ουσίε, όπου έχουμε συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα ΕΕ, για παράδειγμα, με, το πρόγραμμα, με ένα πρόγραμμα για την κοκαίνη και την ηρωίνη και σε ό,τι αφορά τα συνθετικά ναρκωτικά εν γέννη. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνουμε την διαδικασία, όχι μόνο τη διαδικασία για τα αμα, ναρκωτικά, αλλά και για τους προδρόμους ε, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όχι μόνο, δηλαδή, να κοιτάξουμε το τελικό προϊόν. Το ερώτημα που έθεσε η κυρία Σίπελ. Πολλά ερωτήματα κάνατε. Κάποιες βασικές απαντήσεις. Η παραγωγή κάναβης και συνθετικών ναρκωτικών και έκσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και ο συνάδελφος, έχουν ως αποτέλεσμα πολλά απορρίμματα ο κλάδος αυτός έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη παραγωγή απορριμμάτων και αυτές οι χωματερές είναι εντελώς παράνομες στην φύση και συνυπολογίζονται στον αντικτύπο στην, ε, στο περιβάλλον και στην κοινωνία για να καθαρίσουν αυτές οι χωματερές. Πίστεται και το θέμα επιδημιοδολογίας. Ναι, συλλέγουμε λοιπόν τα σχετικά στοιχεία για τα σχετικά λύματα που προκύπτουν και είναι ένα από τα συμπληρωματικά εργαλεία αυτά για να κατανοήσουμε και το πώς αλλάζει η κατανάλωση. Αυτό δεν είναι ένας δείκτης από μόνος τους, αλλά με την ανάλυση πολλαπλών δεικτών σε σχέση και με τις κατασχέσεις και με τα άλλα δεδομένα που έχουμε, μας επιτρέπει να σχηματίσουμε μια συγκεκριμένη εικόνα ακόμα και υπάρξει και πριν υπάρξει σημαντική αύξηση στην κατανάλωση. Για παράδειγμα, έγινε μία ερώτηση για τα συμμετικά ναρκωτικά από διάφορους ευρωβουλευτές να πω ότι πέρσι είχαμε 58 νέες ψυχοτρόπους ουσίες οι οποίες εντοπίστηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά μία κάθε εβδομάδα. Και αυτές είναι οι καινούργιες ουσίες όλες μαζί με αυτέ που έχουν εμφανιστεί δηλαδή τα τελευταία δύο-τρία χρόνια και που κατά καιρού επανεμφανίζονται, μιλάμε για 780 ουσίε. Το 2018 ήταν 370 οι ουσίε οι οποίε επανεμφανίστηκαν στην ευρωπαϊκή αγορά. Τέθηκε το ερώτημα για την ε, τα ποσοστά θανάτων. Το 2018 είχαμε 9.500 θανάτους περίπου ε, ως αποτέλεσμα χρήσης ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Ήταν 72.000 αντίστοιχα ποσά. Μία ερώτηση μου κάνετε για την κάναβη. Έγιναν και κάποιες ερωτήσεις ε, για την κάναβη, τις οποίες θα τις απαντήσω και μετά θα ολοκληρώσω στο σημείο αυτό, γιατί έχετε και την ψηφοφορία σας. Θα ε, σας απαντήσω γραπτά τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Το θέμα της κάναβης, λοιπόν. Καταρχά Αλθεύει το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στο περιεχόμενο στην ισχύ και τη συγκέντρωση των ε, καναβαίδων και στην αστική κάναβη που παράγεται εκτός εντός και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε εμ, στη ε, κάναβης. Στον Καναδά αναφέρθηκε πρόσφατα ότι υπήρξε αύξηση. Αλλά ακόμα δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τον αντικτύπο της αλλαγής της νομοθεσίας στον Καναδά, αλλά φαίνεται ότι αυτό σχετίζεται με το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την κάναβη στη χώρα αυτή. Σε ό,τι αφορά τις ε, ρυθμισμένες αγορές κάναβης, να σας πω μια καλή είδηση οριστικοποιούμε και ολοκληρώνουμε μια σχετική έρευνα που έχει γίνει στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά. Θα την έχουμε σε ένα-δύο μήνες και με χαρά θα σα την παρουσιάσω την έκθεση αυτή όταν θα επιστρέψω. Έχω και πάρα πολλέ άλλε απαντήσει, αλλά θα προτιμούσα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο, για την προσπάθεια που κάνατε και για την ε, προθυμία να δώσετε περαιτέρω στοιχεία γραπτά, γιατί προφανώ ε, τα κράτη-μέλη έχουν εξφράσει έντονο ενδιαφέρον. Η έκθεση του 2019 πραγματικά είναι πολύ ανησυχητική και τα στοιχεία που μας δώσατε επίσης είναι ανησυχητικά. Ναι, και εγώ την ίδια προτίθεμαι να απαντήσω και γραπτά, αν θέλετε, όπως και ο Αλέξης, να σας πω πώς είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ακούσαμε και την προηγούμενη συζήτηση για το πώς ε, θα πρέπει να πάρουμε τα σωστά στοιχεία από τους παρόχους. Αυτό είναι βασικό θέμα. Παγκόσμια πρόσβαση τώρα για τις ε, δυνάμεις ε, εφαρμογής του νόμου. Και εδώ είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Να αναπτύξουμε επίσης ένα νομικό πλαίσιο Η διαδικασία κατάσχεση είναι βασική προπόθεση και η οδηγία για την ξύπλημα χρήματο. Εφαρμόζουμε αυτή τη συνεργασία με τρίτε χώρε και επειδή υπάρχουν μεγάλε αγορέ στην Κεντρική Αμερική θέλουμε πιο στενή συνεργασία με χώρε όπω η Κολομβία με τα κράτη-μέλη, συνεργασία με τον κλάδο. Είδατε από την τελευταία εικόνα του 2020 δεν αγοράζουμε τέτοιο εξοπλισμό προφανώ στους δρόμους. Υπάρχει προφανώς ανάγκη να μιλήσουμε και με το βιομηχανικό κλάδο. Όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν τμήμα μια στρατηγική για το θέμα του λιμάνι, του λιμανιού. Τα τελευταία έξι χρόνια έχουμε αυξήσει και σε ό,τι αφορά τα ποσά που πληρώνονται στου τελωνιακού, τι μπορούμε να κάνουμε για του νέου τώρα. Είναι πραγματικά εύκολο χρήμα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση και θεωρώ ότι τα δεντολογικά εμπόδια, το ηθικό εμπόδιο για να ξεκινήσει κανείς τέτοιου είδου business ε, είναι χαμηλό. Δεν είναι το ίδιο σαν να μιλάμε για διακίνηση ανθρώπων και ε, είναι εύκολο τελικά να ξεκινήσει ένας νέος και να καταλήξει τελικά σε συμμορίες, δολοφονίες κτλ. Να δούμε πόσο συμφετικά ναρκωτικά παράγονται. Βλέπετε κάποια τα στοιχεία στο έγγραφο, αλλά βλέπουμε και πάλι μεγάλη αύξηση κοιτώντας την έκθεση του 2016 και συγκρίνοντας, για τα δεδομένα, τα στοιχεία. Συγγνώμη, λέει ο μιλητής. Για το θέμα της ρύθμισης και του τη νομοθεσία. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών, δεν δικό μα θέμα. Εγώ αυτό που τονίζω είναι ότι δεν υπάρχει ε, μία αγορά σε κάθε χώρα. Είναι παγκόσμια η αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο πλαίσιο. Και με χαρά να απαντήσω ό,τι άλλες ερωτήσει υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ όλα για τις απαντήσεις αυτές οι οποίες πραγματικά ήταν πολύ εύστοχες και αναφέρθηκαν σε πολλές από τις ανησυχίες μας. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό και να διαβάζουμε τις εκθέσει σα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσπάθειές σας για να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό μοντέλο, αυτή η ευρωπαϊκή προσέγγιση. Μου προκαλεί σοκ το γεγονός ότι η σύγκριση των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα ναρκωτικά είναι 9.500 άτομα, ενώ στις ΗΠΑ είναι 72.000 ε, άτομα. Αυτά. Κάτι πρέπει λοιπόν να εξαγάγουμε συμπέρασμα από τόσο υψηλό αριθμό θυμάτων. να ψηφίσουμε και να ευχαριστήσουμε τους ε, δερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, να κάνουμε την ψηφοφορία για την σχέδιο συστασής. Για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σερβίας. Όχι, Σερβία, συγγνώμη, Μαυροβουνίου. Με το Μαυροβούνιο. Για την αρχή την συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Η κυρία Φόλαφ είναι η συγγήτρια. Μία τροπολογία... Κατευθείαν τελική ψηφοφορία είναι μόνο. Όχι, λάθος. Υπάρχει μία τροπολογία. Υπάρχει μία τροπολογία. Uh, η οποία έχει υποβληθεί από την ΚΟΕ, κυρία Ρέγκο, η οποία θα τεθεί σε ψηφοφορία πρώτα. Ψηφίστε λοιπόν για την τροπολογία παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Υπάρχει μία ε, επιπλέον ψήφος του ΕΛΚ και δύο επιπλέον ψήφοι του όχι, μία επιπλέον ψήφος του ΕΛΚ και μία επιπλέον ψήφος της ΓΚΟΕ. Εντάξει, διορθώθηκε το ΕΛΚ, ένας παραπάνω από την ΓΚΟΕ όμως, τέσσερις είναι. Τέσσερις είναι, λέει ο πρόεδρος. Η γραμματεία μας ε, ζητάει από την ΚΟΕ ένας να αφαιρέσει την κάρτα του. Εντάξει τώρα, μπράβο. Είμαστε σωστά. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. με 9 ψήφους υπέρ 44 κατά. Απορρίπτεται η τροπολογία. Και τώρα θα περάσουμε στην ε, τελική ψηφοφορία, ε, έναρξη ψηφοφορίας. Περιμένει ο Πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορίας με 43 ψήφους υπέρ και 9 κατά εγκρίνεται. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο προσχέδιο σύστασης για το ίδιο θέμα. Μάλλον γιατί έχουμε την ίδια κατάσταση. Έχουμε ουσιαστικά μια πρόταση για να ανατραπεί η σύσταση από την ΚΟΕ. Επομένω θα τεθεί πρώτα σε ψηφοφορία η τροπολογία της ΚΟΕ. Τώρα συζητούμε για την Σερβία και ε, τις σχετικές δραστηριότητες της ΣΥΣΜΗ. Ψηφίζουμε πρώτα την τροπολογία της ΚΟΕ. Ψηφίστε παρακαλώ. Είμαστε καλά από πλευρά ε, απαρτία και αριθμών και αντιπροσώπευση. Πέρα ψηφοφορία. 10 υπέρ, 44 κατά. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία λοιπόν για το προσχέδιο σύσταση. Ψηφίστε παρακαλώ. is closed. Πέρα ψηφοφορία. 44 ψήφους υπέρ και 10 κατά εγκρίνεται. Ευχαριστούμε κυρία Φόλαφ, ο πρόεδρος, ευχαριστεί και τους ε, διερμηνείς. Θα επαναλάβουμε τη συνεδρίαση στις 2.30 με την έκθεση του Επιτρόπου Γιώχανσον. Καλή όρεξη. Προσοχή όμως, όχι 3 το απόγευμα, 2.30. Γεια σας.